Good um, Καλημέρα, συναδελφοί, να ξεκινάμε σιγά-σιγά με έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται. Εγκρίνονται και τα πρακτικά τη 20 Σεπτεμβρίου και 8 Μαρτίου. Ωραία. Διερμηνία δεν υπάρχει σε κροατικά, μαλτέζικα και ελληνικά και μετά περνάμε στην έγκριση συστάσεων των συντονιστών. ορισμός εισηγητών. Εγώ, ο ίδιος, θα είμαι εισηγητής ε, για το σχέδιο ψηφίσματος για το Facebook ε, και την Cambridge Analytica. Ο κύριος De ε, θα είναι για, τον κανονισμό, για τους κανονισμούς που θα ισχύουν και στα μη συμμετέχοντα κράτη-μέλη που αφορούν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη 2020-2027 και για την πρόταση κανονισμού για πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη 2021-2027. Κυρία Σκρίπεκ από το ECR για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην Ιρλανδία και για την εφαρμοστική απόφαση σε σχέση με την βάση DNA και με μια άλλη ανταλλαγή δεδομένων ε, για την Κροατία. Ε, εγκρίνει η Επιτροπή. Ωραία. Το τρίτο θέμα έχουμε ένα διορθωτικό στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την διαχείριση μεγάλων στήματων πληροφορικής στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών που τροποποιεί τον κανονισμο 1896 1897-2006 και 776 και ανακαλεί την σχετική απόφαση και ερχόμαστε σε κάτι που αφορά τις πράξεις κατεξιοδότηση στις πράξεις ε, κατ' το σχέδιο συμφωνίας ε, για την περίοδο των ευρωεκλογών και της πράξης κατεξουσιοδότηση έχει εγκριθεί από την Σύνοδο των Πρόεδρων των Επιτροπών και σας κοινοποιήθηκε μέσω του δελτίου της ε, ΛΥΜΠΕ. Το εγχειρίδιο έχει αναθεωρηθεί. Σύμφωνα με την Διοργανική Συμφωνία του 2016. Η αναθεωρημένη αυτή εκδοχή εγκρίθηκε στις 24 Αυγούστου. Στις 24 Σεπτεμβρίου το Κοινοβούλιο έλαβε το σχέδιο αποφάσεως για την επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων από την Ιαπωνία. Αυτό το είπαν όλα τα μέλη της ΛΥΜΠΕ και ενημερώθηκαν μόνο από την γραμματεία. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει κάποια αντίρρηση, ενημερώσει την γραμματεία μέχρι τις 8 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Και θα το δούμε και στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. Και μάλλον τα λέω γρήγορα, για το θέμα της διερμηνίας. Λοιπόν, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες και πρέπει να εγκρίνουμε το διορθωτικό ε, στον ε, κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν ξέρω, μα δεν ακούει και κανείς. Τέλος πάντων, για τα πρακτικά. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έτσι να είμαστε ακριβείς. Οπότε περνάμε τώρα στο σημείο 4. Η χρήση δεδομένων ε, του χρηστών του είναι Facebook από την Cambridge Analytica και το τι σημαίνει αυτό για την προστασία δεδομένων. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Παρουσιάζουμε το σχέδιο ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 123 με το θέμα που σας ανέφερα. Το ψήφισμα βεβαίως προέκυψε μετά από την δουλειά που έγινε μετά από την ακρόαση στην διάσκεψη των Προέδρων αλλά και τρεις άλλες ακροάσεις που οργάνωσε η Επιτροπή μας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, ανεπλάγησαν σε τις ακροάσεις που έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και βεβαίως πρόκειται για κάτι το οποίο είναι λογική συνέχεια των γεγονότων της διαρροής ε, δεδομένων και την κατάχρηση των δεδομένων αυτών. Βεβαίω ε, δεν είναι μόνο η πολιτική και οι δράσεις του Facebook που επηρέασαν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ίσως να επηρέασαν ε, και τα αποτελέσματα εκλογών και την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ψηφιακές πλατφόρμες. Εξ λοιπόν του Προέδρου, όπως ξέρετε, οργανώθηκε μια πρώτη ακρόαση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Facebook, τον κύριο Ζούκερμπερκ, στις 22 Μαΐου και μετά έγιναν και άλλες ακροάσεις από την ΛΥΜΠΕ σε στενή συνεργασία με τις Επιτροπές Ήτρε, και Γιούρι. Λοιπόν, τα ερωτήματα των ε, κρατών μελών και οι απαντήσεις ε, του Facebook ε, και Λοιπόν, απαντήθηκαν από την Εκλογική Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών, με μονομένους δημοσιογράφους, ακτιβιστές, τους αρμόδιους επιτρόπους. Όλοι αυτοί μας ε, έδωσαν απαντήσεις ε, οι οποίες μας βοήθησαν πάρα πολύ και θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκομένους. Λοιπόν, τις τελευταίες αυτές εβδομάδες συνεργάστηκα στενά με επικεφαλής πολιτικών ομάδων για να συντάξουμε το κείμενο που έχουμε μπροστά μας και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ισορροπημένο, σαφές ε, κείμενο και ζητάει από τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να φροντίσουν να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα. Συναδελφοί, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι όταν λέω ότι απογοητευτήκαμε ε, από την απόφαση του Facebook να μην στείλει προσωπικό με την απαραίτητη τεχνική εμπειρία και εταιρική ευθύνη για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, σε έλλειψη πληροφοριών ή σε έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, οπότε προτείνω στο κείμενο να ζητήσουμε έναν ανεξάρτητο έλεγχο του Facebook από την ΕΝΙΣΑ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα. Ζητάμε λοιπόν πλήρη ανεξάρτητο έλεγχο του Facebook από την ΕΝΙΣΑ. Επιπλέον πρέπει να δούμε το πώς τα πολιτικά κόμματα και οι εκστρατείες χρησιμοποιούν τις κοινωνικές πλατφόρμες για τις ε, προεκλογικές εκστρατείες. Ένα κώδικα συμπεριφορά με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων πρέπει να αναπτυχθεί. Αν δεν γίνει αυτό θεωρώ ότι απαιτείται νομοθετική δράση και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάσουν οι βουλευτές. Αλλά συνάδελφοι υπάρχει επίσης το γεγονός ότι οι εταιρείε πρέπει να εφαρμόζουν ε, και να συμμορφώνονται με το GDPR. Και εμείς βεβαίως να προχωρήσουμε με την οδηγία περί ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας. Ε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε την γενική οδηγία και τα είχαμε θέσει αυτά και στον κύριο Ζούκερμπεργκ στην ακρόαση όπου και ο ίδιος είχε πει ότι το GDPR δεν είναι η μόνη ε, συμμόρφωση η οποία απαιτείται. Οπότε πρέπει να δούμε ακριβώς την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα ως το επιπλέον πλαίσιο που απαιτείται σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε με το Facebook. Οπότε ζητώ από το Συμβούλιο να ακούσει αυτά τα αιτήματα περί νομοθετικής δράσης. Οπότε με αυτά τα δεδομένα, αλλά όπως ξέρουμε έχουμε και άλλα δεδομένα, στο ψήφισμα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Να ξεκινήσουν οι συντονιστές, οι παρόντες δηλαδή. Να ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα μιλήσει εξ ονόματος της κυρίας Μετσόλα. Άξελ, έχει τον λόγο αγαπητέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απενός βεβαίως είμαι ικανοποιημένος για το ότι ολοκληρώθηκε αυτή η φάση της έρευνας γιατί είχα την εντύπωση ότι ε, έχουμε κάποιες επαναλήψεις ε, και στις ερωτήσεις και στις διαδικασίες αλλά τέλος πάντων ήταν ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις το ερώτημα σε ποιο βαθμό τώρα ε, χρειάζεται να ξεκινήσει ή αν μπορούμε να κάνουμε μια έρευνα και το αν θα γίνει μέσω της ενίσα είναι κάπως αμφίβολο θεωρώ εγώ γιατί δεν είναι τόσο απλό να εκτιμήσουμε το εάν η ενίσα έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο ε, για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εφενός έχουμε εθνικούς επόπτες δεδομένων ε, Ευρωπαίο επόπτη δεδομένων που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, οπότε δεν είμαι σίγουρος για το εάν η ΕΝΙΖΑ είναι η κατάλληλη ερευνητική αρχή. Και μετά το άλλο είναι το πώς θα περιορίσουμε τελικά μια τέτοια έρευνα. Θα ξεκινήσει που στην Ιρλανδία, στη ΣΥΠΑ, έχουμε κάποια αρμοδιότητα στη ΣΥΠΑ. και σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα περιοριστούμε. και δεν ξέρω καν αν αφορά Ευρωπαίους πολίτες και ποιους Ευρωπαίους πολίτες αφορά. Είναι δύσκολο αυτά να εκτιμηθούν. από νέες ιδέες, νέους ε, κανονισμούς. Δηλαδή, εντάξει, απαγορεύουμε. Απαγορεύουμε και διάφορα πράγματα. Απαγορεύουμε και την απάτη, την κλοπή, ε, τον φόνο, αλλά συμβαίνουν. Αυτό το οποίο θα βοηθήσει είναι η εντονότερη έλεγχη Οπότε λείπει ακριβώς από ε, τη χρονική σκοπιά και η σχετική οδηγία. Ή μάλλον είχε προβληθεί κάπως αργότερα η εφαρμογή της. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο πώς ε, μπορούμε για τέτοιες ε, περιπτώσεις να δράσουμε προληπτικά και να ενισχύσουμε τον έλεγχο. Γιατί αλλιώ δεν βλέπω κάποιο νόημα. Δηλαδή, καταχρήσεις θα υπάρχουν και στο μέλλον. Ε, Αν αρχίζουμε κάθε φορά να δρώμε μέσω της ενίσα, είναι και δυσανάλογο. Γι' αυτό θεωρώ Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν. Πρόκειται για μια κατάχρηση δεδομένων που πρέπει να καταπολεμηθεί, να ελεγχθεί και να δούμε μετά αν υπάρχουν κάποια κένα στην εφαρμογή του σχετικού κανονισμού. Να δούμε δηλαδή αν έχουμε κάποιους επαρκείς σχετικούς ε, μηχανισμούς ε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε κάπου παραπέρα γι' αυτό είμαι κάπως επιφυλακτικός και νομίζω ε, εκεί πρέπει να μείνουμε, δεν είναι να πάμε παραπέρα. Ευχαριστώ, κύριε Βόσο. Στο τέλος, αφού ακούσω όλους τους συναδέλους απαντήσω, αλλά αρχικά μπορώ να πω ήδη ότι τώρα συζητούμε ακριβώς πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί και να δράσει ανησυχίες που προέκυψαν από την υπόθεση αυτή του Facebook εντολή είναι εμείς το Κοινοβούλιο πώς θα ανταποκριθούμε στις ανησυχίε των πολιτών απέναντι στο Facebook. Όλα αυτά είναι πολύ καλά ορισμένα. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ πεπειραμένων συναδέλφων, πολιτικών ομάδων. Όμως, το Κοινοβούλιο θα έχει σαφείς αρμοδιότητες ρυθμιστικές αλλά και ήπιας αντίδρασης. Στο ψήφισμα, το διαβάσει κανεί, ζητάμε για παράδειγμα τον πλήρη ανεξάρτητο έλεγχο από ΕΝΗΣΑ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων. Είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν αυτά. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει. Και μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτόν. Μιλά για την Eurojust και άλλα. Εγώ θέλω άμεση δράση. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πάντως και τώρα κυρία Ζίπελ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ ο Κλοντ. Για να είμαι ειλικρινής, εξεπλάγει κάπως. Χαίρομαι πάντως που το ΕΛΚ, κύριος Φως συγκεκριμένα, αναγνώρισε τη σημασία του κανονισμού για την προστασία και λέει ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος, να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις του κανονισμού και ελπίζω να πιέσουμε όλοι συνολικά ώστε και οι αρμόδιε αρχέ προστασίας δεδομένων αλλά και η συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να γίνει, να υπάρξει ο κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέσα αυτά νέα καθήκοντα. Δεν φαίνεται όμως αυτό αυτονόητα να λειτουργεί στα κράτη-μέλη προς το παρόν. Για τον περισσότερο έλεγχο και ότι δεν χρειαζόμαστε νέα κανόνε. Ε, μακάρι να το έλεγε και για άλλου τομεί το ΕΛΚ αυτό. Γιατί πολύ συχνά ε, και πολύ εύκολα προτείνουν ε, νέα νομοθεσία, νέους κανόνε. Θα ήθελα να επανέλθω στις ε, ακροάσεις για το Facebook που είχαμε εδώ. Είναι γεγονό ότι υπήρξαν πολλές επαναλήψεις ερωτήσει αλλά για ένα βάσιμο λόγο. Γιατί αυτές οι ακροάσεις ε, δημιουργούσαν πάρα πολλές απορίες που δεν έπαιρναν καμία απάντηση. Είχαμε πει ότι με βάση τον παλαιό κανονισμό ε, δεν ε, χρειαζόταν το Facebook να προσέχει κάποια δεδομένα. απάντηση ήταν ναι, νομίζουμε ότι όλα τα κάναμε σωστά. ποιο κανόνα τήρησαν, έπρεπε να το αποδείξουν αυτό. Κατά την άποψή μου τώρα, δεν μιλάμε για τον έλεγχο συγκεκριμένου περιστατικού. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε απαντήσεις από το Facebook, αυτό είναι το ζήτημα. Και πρέπει γενικά να δούμε τελικά το Facebook. Τηρεί κανόνες προστασίας δεδομένων. Και κατά το παρελθόν φαίνεται ότι συγκέντρωνε μαζικά δεδομένα και όποιος ήθελε να τα πάρει τα αγόραζε ή τα έπαιρνε με άλλο τρόπο. Άρα υπήρξε κάθε είδους χειραγώγηση και εκμετάλλευση των στοιχείων και μέχρι και για τις εκλογικούς λόγους ε, που γνωρίζουμε. Αλλά αυτά τα στοιχεία ε, ή τα αποτελέσματα των εκλογών για παράδειγμα. Ποιος τα αγοράζει, ποιος έχει στον κόσμο ε, επιρροή και χρήματα για να επηρεάσει τόσο πολύ. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια ήταν τα συμφέροντα για αυτή τη χειραγώγηση. Και αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό που θέλουμε να συμπληρώσουμε με το Ευρωπαϊκό Αυτό Συμβούλιο Προστασίας και να προσθέσουμε και το ΕΝΙΖΑ. Σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα που θα προκύψουν και στους ελέγχους για το πώς θα επεξεργάσει τα δεδομένα το Facebook. Υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να κατανοήσουμε. Επομένως, η συμμετοχή του ΕΝΙΖΑ νομίζω είναι πραγματικά κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο, ιδίως για τα τεχνικά ζητήματα, αν θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουμε και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια λογική διαδικασία. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη, θέλουμε να το ελέγξουμε αυτό ή τι γίνεται σε άλλα κράτη. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα, όλα μαζί είναι για την Ιρλανδία ή για κάτι άλλο. Ε, δεν με νοιάζει που ξεκίνησε ή τι έγινε, γιατί Υπάρχει ο κανονισμός ε, περί προστασίας δεδομένων. Υπάρχουν πολίτες, ε, οίκοοι κρατών μελών, ε, οι οποίοι πλήγησαν. Και νομίζω πρέπει να συνεργαστούν όλες οι χώρες, όλοι οι αρμόδιες αρχές και πρέπει να συγκεντρωθούν τα δεδομένα από όλους τους αρμόδιους φορείς μέσω του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει ακριβώ πώ θα προχωρήσει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι προπόθεση και μεγάλη πρόκληση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Facebook στη ΣΥΠΑ, υπάρχει η λεγόμενη απόφαση καταλληλότητα ή επάρκεια, adequacy decision. Ε, στην Ευρώπη είδαμε ότι δεν τήρει του κανόνε, όλου του κανόνε το Facebook. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την υποχρέωση που αναλαμβάνει από μόνο του το Facebook, δεν ξέρω αν την ε, Ούτε καν για τη ΣΥΠΑ, πόσο μάλλον για την Ευρώπη. Δεν είμαι σίγουρη ότι το κάνει αυτό το Facebook. Έχω λοιπόν τι αμφιβολίε μου και για το κατά πόσο τηρούνται από το Facebook όλοι οι κανόνε τη ΣΥΠΑ. Τι κανόνε και για σχέση με την προστασία αυτή, το, τη θωράκιση τη ιδιωτικότητα, το privacy shield. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρη διατύπωση σε κάποια σημεία του ήθελα Θα ήθελαν πιο αυστηρή κριτική μας, αλλά εντάξει θα το δεχτώ. Αυτό το κείμενο είναι ένα έγγραφο που πρέπει να βρει ικανοποιημένε όλες τις άλλες πολιτικές ομάδες ε, και νομίζω ότι αν γίνει δεκτό ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα συμβιβασμός. Έχουμε και τις εκλογές που έρχονται. Και αυτό πρέπει να κάνουμε ώστε να τον γρηγορότερα είναι να προβούμε σε απαραίτητου ελέγχου. Ευχαριστώ. Η CR Στίβεν δεν είναι εδώ. Αν έρθει κάποιο από το ECR θα του δώσω το λόγο. Πάω λοιπόν στην Άλντε. Ούτε η κυρία Γκρισμπέκ είναι εδώ. Αλλά είναι η κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για το ψήφισμα. Και θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η Μπρίγκη Τσίπελ, κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Πάντοτε ευνηδιάζομαι με την ε, επιφυλακτικότητα, για να μην πω άρνηση του ΕΛΚ, να εφαρμόσουν τους ευρωπαϊκούς νόμους, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε τον κανονισμό GDPR για την προστασία των δεδομένων, που, για τον οποίο είμαστε περήφανοι και είναι από του καλύτερου κανόνε για προστασία του ιδιωτικού βίου στον κόσμο και τελικά δεν κάνουμε πραγματική προστασία των πολιτών μα στην πράξη. Προστατεύουμε περισσότερο τι αμερικανικέ εταιρείε από του Ευρωπαίου πολίτε. Αν μου επιτρέπετε να είμαι τόσο κοινική. Τρει σύντομε παρατηρήσει. Πρώτον, πρέπει να δούμε την υλοποίηση και την εφαρμογή οριζοντίως διότι έχουμε μια σπίδα προστασίας της ε, ιδιωτικότητας και την τελειότερη νομοθεσία, αλλά η εφαρμογή της είναι κατάπτυστη. Βλέπουμε ότι όταν ε, ο κανονισμός ε, GDPR εφαρμόστηκε, φνηδιάστηκε πολλοί κόσμος από κάποιες από τις απαιτήσει του κανονισμού. Και ήταν απαιτήσει που προϋπήρχαν από την οδηγία. Αυτό δείχνει σε τι βαθμό η οδηγία δεν εφαρμοζόταν. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε κάπως αυστηρότεροι. Η τεχνολογία εξελίσσεται. Και υπάρχουν παρεμβολές, όχι μόνο στον ιδιωτικό μας βίο, αλλά και στην ε, δημοκρατία, όπως είδαμε στην περίπτωση της Cambridge Analytica και του Facebook. Η δεύτερη παρατήρησή μας αφορά την, αφορά την παράγραφο 24 ακριβώς για το θέμα της επιβολής της εφαρμογής. Νομίζω ότι ορθώς προτείνεται η αρχή προστασίας των δεδομένων να ενισχυθεί. Δεν συμφωνώ όμως ότι θα πρέπει αυτό να γίνει με την εισαγωγή κάποιου τέλους στον ε, τομέα της πληροφορικής. Αυτό είναι πρόβλημα των δημοσίων αρχών. Το έχω ήδη προτείνει, Πρόεδρε, να οργανώσουμε ακρόαση, νομίζω έχει προγραμματιστεί για το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς για το θέμα αυτό. Για το κατά πόσον οι εθνικές κυβερνήσεις δίνουν αρκετά ε, κονδύλια στις αρχές προστασίας των δεδομένων για να, προστατεύουν, για, να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, στη δικιά μου τη χώρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει στι άλλε, παίρνουν ε, τουλάχιστον ένα τρίτο λιγότερο από ό,τι χρειάζονται για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά του. Αυτό σημαίνει ότι δεν ε, φροντίζουμε για το GDPR. Τα κράτη-μέλη δεν είναι ταγμένα σε αυτό το σκοπό. Δεν καλύπτουν τι απαιτήσει. Θα πρέπει να ξεκινήσει με παραβάση διαδικασίε η Επιτροπή. Όχι περισσότερου φόρου ή τέλη. Ο εθνικό προπολογισμό έπρεπε να καλύπτει αυτέ τι αρχέ για τους εθνικούς επόπτες των δεδομένων. Αντί λοιπόν για επιπλέον τέλη, θα έπρεπε να πιέσουμε τις εθνικές αρχές να κάνουν αυτό που οφείλουν. Και τελευταία παρατήρηση, παράγραφοι 25 και 26 για την ασπίδα της ιδιωτικότητας. Έχουμε περάσει ψήφισμα στις 5 Ιουλίου, όπου λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με αυτή την ασπίδα ιδιωτικότητα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Κατά τι δικέ μου πληροφορίε δεν έχει συμβεί απολύτω τίποτα ακόμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια επιπλέον παραγραφό που να λέει ότι ζητούμε την αναστολή τη ασπίδα. Παρόλο που δεν θεωρώ ότι νομικός ε, στέκει αυτό, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ή θα περνάμε νομοθεσία που τόσο πολύ προβάλλεται, κάνουμε τόσο θόρυβο και φασαρία και τι γιορτάζουμε. Και μετά όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση και επιβολή δεν θα γίνει τίποτα. Θα το περνάμε στον τούκου. Προτείνω λοιπόν την συμπερίληψη μιας παραγράφου όχι μόνο για την εισαγωγή, για την έγκριση του ψηφίσματος τον Ιούλιο, να μην μιλάει μόνο γι' αυτό, αλλά να προβλέπει και μια προθεσμία. Και να υπάρξει αναστολή της ασπίδας ιδιωτικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή, και θα το πω με θετικό τρόπο, θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρότερη ε, και αυστηρότερη στην επιβολή. Και πραγματικά τονίζω εδώ το πολύ. Πρόεδρος, για την υλοποίηση και την επιβολή θα ακούσουμε και τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς ε, θα μπορούσε αυτό να καλυφθεί στο πλαίσιο του ψηφίσματος. Ευχαριστούμε Σόφη. Από την ΚΟΕ υπάρχει κανείς. Παρακαλώ, εάν οι συνάδελφοι έρθουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, να ζητήσουν το λόγο. Ο κύριος Ράνης του Ευχαριστώ κύριε Μωρές. Το σκάνδαλο αυτό Facebook Cambridge Analytica δεν είναι μόνο θέμα προστασίας δεδομένων. Είναι σκάνδαλο δημοκρατίας. Έχουμε μια εταιρεία λέγοντας ότι θα κάνει απλώς έρευνα, έλαβε τα δεδομένα 70 εκατομμυρίων χρηστών για να ασκήσει στοχευμένη επιρροή τουλάχιστον στις ΗΠΑ και στο Brexit και υποθέτουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Παρά την ακρόαση που κάναμε, πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά. Πόσα δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών πραγματικά υπέστησαν καταχριστό Το Facebook μας λέει 72 εκατομμύρια και μετά κάνει τελείως στροφή και λέει δεν αφορούν κανένα πολίτη της Ένωσης. Πώς ακριβώς χρησιμοποίησε η Cambridge Analytica τα δεδομένα, με ποιον στόχο και πώς α, ε, μετά παρακίνησε κάποιους ανθρώπους ε, είτε να ψηφίσουν συγκεκριμένη παράταξη είτε να μην πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την παρακολούθηση του θέματος, αλλά βεβαίως το δυσκολότερο θέμα είναι ακριβώς πώς επηρεάζουν όλα αυτά την δημοκρατία μας. Έχουμε πραγματικά ένα φαινόμενο στο οποίο οφείλεται το Brexit και η εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ. Μια ομάδα ερευνητών του Warwick είδε το τι γίνεται στην ε, Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς και κοίταξε κατά τόπους αν σχετίζεται με την ανεργία, την παρουσία αλλοδαπών κτλ. κτλ. Η μοναδική παράμετρος η οποία ήταν σημαντικά διαφορετική ήταν η χρήση του Facebook. Το Facebook είναι λοιπόν πρόβλημα για τη δημοκρατία μας και χωρίς την Cambridge Analytica. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα. Και καλό είναι το ότι το Facebook παραδέχτηκε το ότι θα δώσει τα στοιχεία αυτά στην διάθεση των πανεπιστημιακών. Και βεβαίως υπάρχει και σχετική έρευνα της Ομοσπονδιακής έρευνας, ε, Επιτροπής Εμπορίου της είπαμε συγχωρείτε. αν δούμε παραδείγματο χάρη και ένα άλλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο με τις εκπομπέ. Εάν είχα εγώ να επιλέξω ω καταναλωτή μεταξυ μεταξύ δύο-τριών εταιριών, τι θα έκανα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε διασυνοριακούς κανόνες για έρευνα και για εκπομπές που λένε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν η στοχευμένη πολιτική διαφήμιση με βάση το προφίλ να απαγορευτεί εντελώς. Ναι. Υπάρχουν ήδη επίσης και άλλα φαινόμενα όπως οι διαφορετικές τιμές που επιβάλλονται κτλ. ένα κίνδυνος που δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Δεν είναι δυνατόν τυπικός να συνεχίσουμε να έχουμε εκλογές αλλά το facebook να επιβάλλει τα αποτελέσματα που θέλει και να διαλέγει ποιος θα βλέπει ποιες πληροφορίες και ακριβώ θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα εάν είναι να κάνουμε κάτι πριν τις ευρωεκλογέ. Βεβαίω το ψήφισμα μιλάει κυρίως για διαφάνεια και αυτορύθμιση Σας ευχαριστώ. Πράγματι εδώ μας υπενθυμίσατε το εύρος των ζητημάτων και το ότι πράγματι ο κόσμος αναμένει κάποια δράση από το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, ε, είπα ότι αν εμφανιστεί κανείς θα του δώσω τον λόγο. Δεν ξέρω λοιπόν αν θέλει να μιλήσει κάποιος για το ECR. Ο Νταν Τόλτον, ευχαριστώ, συγγνώμη. Αλλά ψηφιζόταν στην ΕΜΚΟ μια από μου. Η ECR ε, είδε με αποτροπιασμό ε, τη χρήση των στοιχείων από την Cambridge Analytica. Στηρίζουμε τις έρευνες και πιστεύουμε και εμείς ότι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Ο κανονισμός ε, για τα δεδομένα είναι χρήση. Ε, νομοθέτημα το στηρίξαμε. Χαιρόμαστε που έκλεισε και Analytica, που η Βρετανική Επιτροπή ερευνά εντελεχώς ε, και επίσης φαίνεται και το Facebook να έχει καλύτερη συνεργασία με τις Ιρλανδικές Αρχές Προστασίας ε, των και, και με άλλες χώρες. Ε, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη και σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων αυτό το γραφείο ε, να, στις, στο Βασίλειο να έχει καλές σχέσεις με τις ευρωπαϊκές αρχές για την ε, συγκέντρωση σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Για το σχέδιο ψηφίσματος είναι αρκετά μετρημένο. Βέβαια, μας, ε, κάποια από αυτά θεωρούμε που λέγονται ότι είναι υπερβολικά. Υπάρχουν αναφορές που δεν βοηθούν ε, στο Brexit. Υποχρεωτικό σύστημα, δακτυλοσκόπηση για ηλεκτρονική ε, καταγραφή κτλ. Πρέπει να τα δούμε. Είναι και εκτός της Ευρωπαϊκής Αρμοδιότητας. Πάραφος νέα Για το profiling. Ότι απογορεύεται. Δεν ισχύει αυτό. Στο 9 επιτρέπεται. Αλλά υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις από το λόγου. Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων πάνω. Θα μπορούσε λοιπόν να ληφθεί υπόψη το 9 στη διατύπωση Στο 17. Ότι πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο του Facebook λένε. Δεν το αποφασίσουμε στο κοινοβούλιο. Το Facebook θα αποφασίσει ποιο επιχειρηματικό μοντέλο θα ακολουθήσει. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί βέβαια από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη-μέλη. Πρέπει να αλλάξει το 17 και συγκεκριμένα το συγκεκριμένο σημείο διαγραφή. 24. Νέο φόρο για τι πλατφόρμε προβλέπεται. Δεν είναι σωστό χώρο για τη συζήτηση νέων φόρων. Πρέπει να διαγραφεί και αυτή η παράγραφο. Και τέλο, παράγραφο 30, που ζητά από το Συμβούλιο να συνεχίσει το έργο του για το e-privacy. Πρώτον, το GDPR θέλουμε να αρχίσει να ισχύει, να περάσει λίγο χρόνο και μετά να δούμε, αφού το αξιολογήσουμε, αν θα αποφασίσουμε ότι χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία ή όχι. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη στιγμή την παράγραφο 30. Θα συνεχίσουμε όμως να συνεργαζόμαστε με τους άλλους συναδέλφους. Thank you thanks, Σε ευχαριστώ, Νταν. Μπυρκίτ, για διαδικαστικό. Έθελες το λόγο. Ναι, σύντομη παρατήρηση. Νταν, μίλησε για το e-privacy. Θέλω να τονίσω ότι δεν πρόκειται για προσθήκη στο κανονισμό το γενικό. Το GDPR αφορά την προστασία των δεδομένων. Το e-privacy είναι κάτι διαφορετικό. Είναι για την προστασία των επικοινωνιών. Πιο σημαντικό ακόμη. Δεν θα στήριζα λοιπόν την ιδέα ότι αυτό είναι μια προσθήκη που μπορούμε να το ε, προσθέσουμε, να μην το προσθέσουμε το σημείο αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οποιαδήποτε αξιολόγηση του κανονισμού προστασία δεδομένων δεν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται προστασία των επικοινωνιών. Για να το ξεκαθαρίσω αυτό, πρόεδρος. Μάλιστα. Ενημερωτικά. Δεν γνωρίζω τον κανόνα. Αλλά επειδή το είπατε πάρα πολύ ευγενικά, Μπίρκιτ, παρότι δεν το διαδικαστικό, ελπίζω ότι το έλεγε υπόψη ο Ντάν. Η Εκομισιόν. Α, όχι, πριν δώσω το λόγο, υπάρχει άλλος ένας που θέλει το λόγο και μετά η Κομισιόν για να υπάρχει μεγαλύτερη τάξη. Δεν θα ήταν ε, καλό να λάβατε πρόταση το λόγο και να ξανάδινα το λόγο στη, στα μέλη της Επιτροπής. Η Άννα Γκόμες λοιπόν, αλλά σύντομα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε η Πύρκη Τσίπελ, που εκ μέρου τη δική μου πολιτική ομάδα. Θα ήθελα όμω. συγκεκριμένα να στηρίξω αυτά που λέει η 24, ανάγκη φορολογίας. Η φορολογία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και για να μειώσει τη δύναμη εταιρεών όπως το Facebook, αλλά και για να παράσχει πόρους και μέσα για τις αρχές μας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να μπορέσουν να στελεχωθούν, να εξοπλιστούν οι ρυθμιστές, ε, οι επόπτες και όλοι αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους ώστε να είναι σεβαστές οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Το πρόβλημα, το είπε και η Σοφ είναι το εξή. Πάρα πολύ ωραίο είναι ο Γενικό Κανονισμό, αλλά δεν δίνουμε δεκάρα για την εφαρμογή του και την επιβολή του. Μεταξύ άλλων, διότι δεν έχουμε ανθρώπους ε, με το σωστό εξοπλισμό που να δουλεύουν ε, εθνικοί επόπτες, προστασίες δομών κτλ. Ε, στις απαραίτητες υπηρεσίες λοιπόν δεν έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό ή την κατάλληλη στελέχωση. Ένας τομέας που πιστεύω ότι πρέπει να περιληφθεί στο ψήφισμα είναι κάτι που προέκυψε από τις δικές μας έρευνες. Η διασύνδεση Cambridge αναλυτικά και Facebook. Ενώ το ότι έδωσε στην Cambridge Analytica τα στοιχεία το Facebook. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Μιλάμε για παραβίαση ε, της ιδιωτικότητας των δεδομένων των πολιτών και φάνηκε τελικά ότι αυτός θα ήταν ένας τρόπος που θα έδινε τη δυνατότητα και στο οργανωμένο έγκλημα να δράσει και να δει στις χώρες μας. Cambridge Analytica και SEL. Είχα μια σχέση. Η SEL σχετίζεται με χώρες που πουλάνε διαβατήρια, που πουλάνε υπηκότητα. ήταν ένα σύστημα στοχευμένο που θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν οι κλιματικές οργανώσεις. Μην το παραβλέψουμε αυτό. Τέλος, να πω. Φυσικά και μιλάμε τώρα για το σκάνδαλο Facebook και Cambridge Analytica, αλλά αν θέλουμε σοβαρά ε, να πάρουμε ε, τα θέματα της προστασίας ε, των δεδομένων, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και αυτά τα οποία γίνονται με τις κινέζικες εταιρείες που είναι ήδη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν συνάψει συμβάσεις με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για το χάρη συστήματα αναγνώριση ε, χαρακτηριστικών του προσώπου πολιτών. Η Huawei, Huawei για παράδειγμα. Και στην Κίνα τώρα έχουν ένα σύστημα που λέγεται Personal Scorecard και κάνει αναγνώριση προσώπου, τεχνητή νοημοσύνη και ελέγχονται όλοι οι πολίτες με αυτόν τον τρόπο. Αυτό εντάξει αφορά προς το παρόν την κινέζικη κοινωνία μέχρι το 2023 θα έχει εφαρμοστεί πλήρω. Τυχαίο όμως είναι ότι ήδη δραστηριοποιούνται σε χώρε μέλη τη Ένωση με τις κάμερες κλειστού ε, κυκλώματος τηλεόραση και χρησιμοποιούν την ε, την νοημοσύνη. Πρέπει να το... Ναι, ναι, ναι, Άννα, ε, Λέω πρόσωπο. Πρέπει να δούμε τι κάνουν και, και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι, Άννα, ναι, Άννα. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται στα κρατημέρια. Ναι, Άννα, ναι, Άννα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα και την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια είναι ότι οι των τελευταίων μηνών για το Facebook και την Cambridge Analytica έδειξαν ανάγλυφα πώς οι εταιρείε χειρίζονται τα δεδομένα των πολιτών και πώς συνολικά εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνες του GDPR. Αυτό που σήμερα συζητούμε. Η όλη υπόθεση δημιούργησε ανησυχίες και για τις ελεύθερες και ανεξάρτητες εκλογές. Προηγουμένως το θεωρούσαμε δεδομένο αυτό. Τώρα όμως δεν ισχύει. Αυτό ήταν μια κλίση για να ξυπνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Το 2019 λοιπόν είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι για το θέμα και το τόνισε και ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης. Καλωσορίζουμε λοιπόν το σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και στρεφόμαστε κυρίως στα προκαταρκτικά πορίσματα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του ΙΒ για την υπόθεση αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις ε, συμφωνούμε με όσα αναφέρει το δικό σας ψήφισμα. Χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση. Για την περίπτωση του Facebook, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε στενή επαφή με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασία Δεδομένων, Word, και τον ομόλογο στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι επικεφαλής της έρευνας αυτής για την Cambridge Analytica. Και καλωσορίζουμε τη συλλογική απόκριση για τις αρχές αυτές. Η Επίτροπος Γιούροβα παρακολούθησε με προσοχή τα πορίσματα της έρευνας και ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες για την υπόθεση. Άλλωστε, προσεχώ θα έχουμε και τη δεύτερη ετήσια αναθεώρηση τη ασπίδα ιδιωτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει την επιβολή πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν αστειευόμαστε με αυτά. Το έχετε δει αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις πολιτικές ε, υποθέσεις που είχαν ε, και πολλές λεπτές προεκτάσεις και πώς ασχοληθήκαμε με αυτές. Το Facebook βέβαια είναι ένα περιπλοκότερο πρόβλημα. Παρελαμβάνεται ένα φάσμα αρχών, πολιτικών κομμάτων, εταιριών που αναλύουν δεδομένα, όσων πουλάνε τα δεδομένα ως ενδιάμεση. Δεν μπορεί λοιπόν ε, οι αρχές να λειτουργούν μεμονωμένα ε, κάθε μια μόνη της. Πρέπει να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να προστατεύσουμε τις εκλογικέ διαδικασίες στην Ευρώπη. Η υπόθεση άπτεται και της ε, πολιτικής διαφήμισης και του ποιο την κοινή. Οι πολίτες πώς γίνονται στόχος. Η ιδιωτικότητα και η κυβερνοασφάλεια πώς εξασφαλίζονται. Ε, για να αναφέρω μόνο μερικέ μέρημνε. Χρειάζεται λοιπόν μια σφαιρική προσέγγιση, ώστε όλε οι αρχέ που ασχολούνται με τα θέματα αυτά να ενώσουν τι προσπάθειέ του. Αυτό στόχευε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πακέτο για του εκλογικού νόμου που προτείναμε στι 12 Σεπτεμβρίου. Λίγα λόγια για το περιεχόμενο του πακέτου. Τρία στοιχεία Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εκλογικές αρχές, οι αρχές προστασία δεδομένων και οι αρχές κυβερνοασφάλεια συνεργάζονται και ανοιχνεύουν που υπάρχουν προβλήματα, συντονίζουν την επιβολή των ισχυρών των κανόνων και εντοπίζουν ελλείψεις και κενά. Στη σύστασή μα ε, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να οργανώσουν δείκτε σε εθνικό επίπεδο για το σκοπό αυτό. Επίση, απευθύνουμε έκκληση να προσαρμόσουν του εκλογικού του κανόνε, ε, μεταξύ των οποίων τη διαδικτυακή ε, προεκλογική εκστατεία και την διαφήμιση ώστε να γνωρίζουμε την χρηματοδότηση, ποιο πλήρωσε την περίοδο αποσιώπηση και ούτω καθεξής για να υπάρχουν σαφεί κανόνε για όλου στις εκλογές του 2019 θα έχουμε για πρώτη φορά εφαρμογή των κανόνων αυτών, των νέων κανόνων. Γι' αυτό οι εκλογικές αρχές και οι άλλοι υπεύθυνοι φορείς θα πρέπει κατεπηγόντως να κοιτάξουν κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Έχουμε λοιπόν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για αυτούς ως μέρος του πακέτου. Τρίτον, Έχουμε προτείνει και νομοθετική τροπολογία αναθεώρηση ε, του κανονισμού 1141 ε, του 2014 για να ελέγξουμε και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Στόχος της τροπολογίας ή αυτή είναι να μπορέσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα να ε, επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων προστασίας της ιδιωτικότητας με σκοπό σκοπίμως να επηρεαστούν τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Τα πρόστιμα θα φτάνουν το 5% του εθνικού προπολογισμού ε, ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος. Ο στόχος είναι όλα αυτά να υλοποιηθούν και να επιβληθούν αποτελεσματικά μέχρι τις εκλογές του 19. Γι' αυτό παροτρύνουμε τους νομοθέτες να ε, προχωρήσουν αμελητή. Ολοκληρώνοντα, θα συνεργαστούμε με το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του ερχόμενου μήνε για να βεβαιωθούμε ότι θα πετύχει η ε, εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η διάσκεψη ψηλού επίπεδου που πρότεινε ο Επίτροπο Κίνγκ για τις κυβερνοαπειλές κατά των εκλογών τον Οκτώβριο θα είναι η επόμενη φάση, καθώ και η μερίδα για τα εκλογικά δικαιώματα στο τέλη Νοεμβρίου. Εκεί θα παραστούν και η Επιτροπή Γιούροβα και ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαν. Τους επόμενους μήνες πρωτού γίνουν οι ευρωεκλογέ, θα περάσουμε ένα διάστημα κρίσιμη σημασία. Θα ζητούσα λοιπόν από το Κοινοβούλιο στο σχέδιο ψηφίσματό του να ευαισθητοποιήσει όλου του ενδιαφερόμενου φορεί για να έχουμε ελεύθερε και ανεξάρτητε και δίκαιε εκλογέ και να προστατευτούν τα δικαιώματα των πολιτών. Thank you very much. Still... Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, οι περισσότερες πολιτικές ομάδες μίλησαν. Ε, υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Εάν όχι, να σας πω ότι για να ψηφίσουμε στις 10 Οκτωβρίου, ε, να πάει στην Ολομέλεια τη 2η του Οκτωβρίου, η προθεσμία είναι αύριο στις 6 ώρα ακριβώς για τροπολογίες. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και ε, σας ευχαριστώ και σας. Ε, περνάμε τώρα σημείο 5. Η κατάσταση ε, περί επάρκειας ε, της Ιαπωνίας. Ποιος έχουμε εδώ, αντικαταστάθηκε ο κύριος, μάλιστα. Δεν έχει έρθει. Τι να κάνουμε, ρε. Um, ναι, ναι, δεν έχει έρθει ο συνάδελφος. Ανά πάσα στιγμή καταπλέει με θορμίσα καθέκτου, με ειδοποιούν. Okay.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 Colleagues, we're going to hear the Commission's representative is going to update the committee on the state of play on the negotiations between the Commission and Japan. Έχουμε λοιπόν τώρα το θέμα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα και την επάρκεια προστασίας από την Ιαπωνία. Την προηγούμενη εβδομάδα λάβαμε κάποια έγγραφα που έστειλε η Κομισιόν και τα προωθήσαμε στους βουλευτές και τους βουλευτές βεβαίως που είχαν πάει και στην Ιαπωνία προσφάτως. Οπότε ο κύριος Τζενκαρέλη έχει τον λόγο για 10 λεπτά το πολύ για να μας ενημερώσει για την αξιολόγηση αυτή. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να με συγχωρείτε. Ε, μου παίρνει 10 η ώρα και εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Όπως θα θυμάστε, τον Ιούλιο που μας πέρασε ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Μου είπα να είμαι σύντομος, λοιπόν θα μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα. Αφενός να τονίσω την ε, σημασία της ε, απόφασης αυτής ε, και της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων και ταυτόχρονα βεβαίως να τονίσω το, τα στοιχεία αυτής της απόφασης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, πιθανώς η πιο σημαντική που προτείνουμε, για μια σειρά διαφορετικών λόγων. Να αναφέρω κάποιους από αυτούς. Πρώτα απ' όλα, εάν εγκριθεί η απόφαση αυτή θα αυξήσει την προστασία των υποκειμένων δεδομένων σε έναν από τους κυριότερους ε, πολιτικούς και εμπορικούς εταίρους με, τον οποίο ήδη σήμερα έχουμε πολλές ανταλλαγές δεδομένων. Αυτή η απόφαση επίση δείχνει, αν μου επιτρέπετε, πως η σύγκληση όταν μιλάμε για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων αποδίδει. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία προσφάτως το Μάιο του 2017, φαίνεται ότι ο Μάιος είναι ο μήνας της ιδιωτικότητας, μεταρρύθμισε τη σχετική νομοθεσία. με βάση μια παρόμοια δομή και διασφαλίσεις ε, και εποπτεία ακριβώς έχει ανεξάρτητες αρχές ε, προστασίας ε, δεδομένων κάτι το οποίο είναι πολύ παρόμοιο με το δικό μας σύστημα. Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, είναι κάτι το οποίο ξέρετε, το είδατε ο ίδιος κατά την ε, επίσκεψή σας ε, στην Ιαπωνία. Και βεβαίως ε, αναγνωρίζοντας αυτόν τον σημαντικό βαθμό σύγκλησης είναι κάτι το οποίο στέλνει και ένα σημαντικό μήνυμα σε άλλες χώρες από την Χιλή και τη Βραζιλία μέχρι την Νέα Κορέα και την Ινδία την Νότια Κορέα και την Ινδία κατόπιν το θέμα αυτής της διαδικασίας επάρκειας, όπως λέγεται, που όπως ξέρετε πάει παράλληλα με την διαδικασία στρατηγικής οικονομικής ε, συνεργασίας ε, ε, οδήγησε σε μια επιτάχυνση της διαδικασίας επάρκειας και η διπλή μας αυτή προσέγγιση είναι η σωστή. Και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό μήνυμα και σε άλλους εταίρους μας. Τι εννοώ δηλαδή. Εννοώ ότι προωθώντας ε, υψηλά επίπεδα προστασίας δεδομένων και, ενισχύ, και το να ενισχύσουμε το εμπόριο δεν είναι πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα. Αντιθέτως θα έλεγα. Και όπως έχετε πει ήδη πολλές φορές, εμείς θεωρούμε ότι η ιδιωτικότητα είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Και ακριβώ επειδή υπάρχει αυτός ο μεγάλος βαθμός σύγκλησης, μπορούμε να ε, συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε τα ωφέλη της εμπορικής συμφωνίας. Και μάλιστα για πρώτη φορά υπάρχει μια αμοιβαία αναγνώριση αμφίπλευρη. Έχουμε λοιπόν ελεύθερες και ασφαλείς ε, ροές ε, δεδομένων και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Σημαντικό αυτό για τις επιχειρήσεις, ε, για την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ως μήνυμα το οποίο στέλνουμε. Γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε και άλλες περιοχές στον κόσμο που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για αυτά τα ζητήματα και το επίπεδο προστασίας. Τώρα όσον αφορά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων έχετε δει ότι έχουμε πολύ εκτεταμένο προσχέδιο με σημαντικά παραρτήματα θα έχετε δει τις λεπτομέρειες απλά να αναφέρω το εξής Καθώς υπάρχει σημαντικός βαθμός σύγκλησης, διαπραγματευτήκαμε και κάποιες επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύσουμε ακριβώς καλύτερα την μεταφορά δεδομένων στην Ιαπωνία. Και βέβαια, ε, όσον αφορά και την ε, πρόσβαση από τις Ιαπωνικές αρχές στα δεδομένα. Να αναφέρω τρία σημαντικά ζητήματα Πρώτα απ' όλα διαπραγματευτήκαμε κάποιους κανόνες που παρέχουν ε, στα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες επιπλέον διασφαλίσεις για τις διαφορές που είδαμε μεταξύ του Ιαπωνικού και του Ευρωπαϊκού συστήματος. Οι επιπλέον αυτές διασφαλίσεις αφορούν παραδείγματος χάρη την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και αυτό δεν ήταν προφανές ή εύκολο. Ευθυγραμμίσαμε τον ορισμό των ευαίσθητων δεδομένων και βεβαίως οι διασφαλίσεις αφορούν και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να μεταφερθούν τα δεδομένα αυτά εκτός Ιαπωνία σε τρίτη χώρα οι λεγόμενες περαιτέρω μεταφορές. Έχουμε και άλλες διασφαλίσεις όσον αφορά την άσκηση ατομικών δικαιωμάτων πρόσβασης ε, στα δεδομένα. Και υπάρχει ακριβώς και η έννοια των ανώνυμων δεδομένων, η διαχωριστική γραμμή της ε, νομοθεσίας ε, προσωπικών δεδομένων και όσων θεωρούνται πλέον ανώνυμα και άρα πλέον δεν προστατεύονται αυτά μιλάμε για ανώνυμα δεδομένα, εννοούμε το ίδιο πράγμα και στις δύο πλευρές. Ε, δεδομένα τα οποία ε, πλέον δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν και αυτό έχει γίνει με τρόπο αμετάκλητο. Οπότε έχουμε τους κανόνες και το πρώτο παράρτημα. Αυτά θα είναι δεσμευτικά για τις ιαπωνικές εταιρείε που εισάγουν δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως θα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε πλήρως ε, και σε σχέση με την Ιαπωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και στα δικαστήρια. Δεύτερη πτυχή, ε, λάβαμε κάποιες διαβεβαιώσεις από τα υψηλότερα κλιμακιά, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υφυπουργό Άμυνας για τον περιορισμό όσον αφορά την πρόσβαση από τις Ιαπωνικές αρχές, τις αστυνομικές αρχές, ε, τις αρχές εθνικής ασφαλείας, στα δεδομένα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιαπωνία, διασφαλίσεις ε, που αφορούν ουσιαστικά το ότι όταν θα υπάρχει πρόσβαση θα υπάρχουν και θα ισχύουν οι αρχές της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας και θα υπάρχει ένας μηχανισμός πρόσφυγης. Βεβαίως να τονίσω ότι η Ιαπωνία όπως οποιοδήποτε σύγχρονο σύστημα στον κόσμο ε, έχει να αντιμετωπίσει και κάποιες απειλές ε, στην ε, περιοχή της και βεβαίως υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο εθνικής ασφαλείας για ιστορικούς λόγους ε, που σχετίζονται με το μεταπολεμικό σύνταγμα της Ιαπωνίας. Και παίζει κεντρικό ρόλο ακριβώς ε, το δικαστήριο το οποίο πρέπει να εκδώσει κάποιο ένταλμα πριν την πρόσβαση στα δεδομένα. Τέλος υπάρχει ένας μηχανισμός ε, προσφυγών για την επίλυση των προσφυγών. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον νέο μηχανισμό που θα φτάνει μέχρι και την διαγραφή των δεδομένων εάν ε, υπάρχει κάποια παράνομη πρόσβαση σε αυτά. Και βεβαίως ε, εποπτεία και διαχείριση θα έχει η Ιαπωνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων πλήρως ανεξάρτητη. Να κλείσω λέγοντας ότι όταν κάναμε την αξιολόγησή μας και διαπραγματευόμασταν ε, τις ε, δικλίδες αυτές ε, παρακολουθούσαμε στενά και τον κατάλογο την ε, λίστα ε, που όρισε ο Ευρωπαίος ε, επόπτης προσωπικών δεδομένων για να δούμε ακριβώς το επίπεδο επάρκειας της ισοδυναμίας. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο θέμα. Έχουμε τον Ευρωπαίο Επόπτη Δεδομένων και όπως γνωρίζετε η απόφαση αυτή έχει τώρα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που θα την εξετάσει τους επόμενους μήνες και αυτό είναι το πρώτο βήμα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνει μετά την διαδικασία της επιτροπολογίας πριν μπορέσει να εγκρίνει το σώμα των επιτροπών. Ελπίζω μην ξεπέρασα τα 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Αναμένω την συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, και Τζανκαρέλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή. Και ήταν και παραγωγική, γιατί είχαμε και τις ε, συνομιλίες για την εταιρική σχέση παράλληλα. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ για να πάρει το λόγο. Να ελέγξω κάτι. Αν είπατε αυτά που ήθελα εγώ ε, τα είπατε, αλλά είναι ένα που δεν το είπατε. Ένα από τα επίμαχα ζητήματα. της μη επίσημης μετάφρασης ε, της ιαπωνικής ε, νομοθετικής πράξης για την προστασία των δεδομένων. Νομίζω ότι ό,τι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει μεταφραστεί ο σχετικός νόμος αλλά δεν υπάρχει ε, νομο... δεν υπήρξε νομοτεχνικός έλεγχος, δεν ελέγχθηκε από αγγλόφωνο νομομαθή, λέει το δικαστήριο αυτό, ο νόμος. Αν μπορείτε να μας διευκρινίσετε. Πώς εγκρίθηκε αυτή η απόφαση, το σχέδιο απόφασης. Αν δεν υπάρχει επίσημη νομική μετάφραση, τι θα γίνει με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Το θέσαμε τότε που πήγαμε εκεί. Δώστε μας και κάποιο ε, χρονοδιάγραμμα όταν θα εγκριθεί απόφαση. Έχουμε και κάποιους ε, Ιάπωνες, ε, τους οποίους και καλώς εδώ. Κυρία Σίπελ και Άννα και ο κύριος Ντάλτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ξέρουμε ότι οι συμφωνίες ε, καταλληλότητας είναι δύσκολες. Θα επικεντρωθώ σε δύο-τρία ερωτήματα είδα ότι υπάρχουν πρόσθετοι κανόνες στο παράρτημα 1. Υποτίθεται ότι θα είναι δεσμευτικοί για τι ιαπωνικέ εταιρείε. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε όμως για τη νομική δεσμευτικότητα των κανόνων. Τέλο ποια θα είναι η νομική του ε, το νομικό καθεστώς. Και φαίνεται ότι θα, θα αφορούν μόνο τα δεδομένα των ευρωπαϊκών πολιτών, όχι των Ιαπώνων ή δεδομένα άλλων χωρών, άλλων δικαιοδοσιών. Τι θα γίνει δηλαδή με τα, την προστασία των δικαιωμάτων των άλλων πολιτών. Και αυτό πώς ευθυγραμμίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και με το, αυτό, αυτό που έχει απαιτήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να υπάρχει ένα επαρκέ επίπεδο προστασία των δεδομένων και σε τρίτε χώρε. Ένα άλλο θέμα που το συζητούμε και το ξανασυζητούμε είναι τα πρόστιμα. 300.000 γεν έως 1 εκατομμύριο γεν. 2.300 ευρώ δηλαδή έως 7.500 ε, και κάτι ευρώ. Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είχαμε συζητήσει το θέμα και είχαμε πει ότι υπάρχει ένα ε, ε, θέμα, υπάρχει μια πολιτιστική διαφορά. Δεν είναι η ίδια για το χρήμα, αλλά είναι ανοίξει στον πολιτισμένο κόσμο η Ιαπωνία. Και δίνεται εντύπωση ότι στην Ιαπωνία η παραβίαση των δεδομένων και της προστασίας τους δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αυτό πώ θα ευθυγραμμιστεί με την απέτηση του Γενικού Κανονισμού ότι περνάνε αποτελεσματικέ, ε, συγγνώμη, αναλογικέ και αποτρεπτικέ οι ποινέ και τα πρόστιμα. Αυτά. Ναι, πράγματι, θα τα πει και ο κύριο Ντάλτον. Πολλά συζητήσαμε σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα. Είναι τέλειως διαφορετικό το καθεστώς στην Ιαπωνία. Έγιναν πολλές φιλοσοφικές συζητήσεις από αυτού, πολύ ενδιαφέρουσες. Τα είπαμε και με τους Ιάπωνες συνομιλητές. Νταν, για πέστα μας τώρα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ναι, τα πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή αυτή στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες ε, ε, πραγματικά σωστά είναι υπερήφανοι με τους κανόνες ε, προστασίας δεδομένων τους. Θεωρούσαν ότι είναι πολύ κοντά σε εμά. Τα ίδια πρόθεση έχουν και Νομίζω αυτό φαίνεται και από αυτά που είπατε εσείς. Μια ερώτηση σε σχέση με κάτι από αυτά που είπατε για την σχέση αυτή που έχουμε μεταξύ μας. Μεταξύ Απονής και Σένους. Και πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό άλλους εταίρους. Γιατί εγώ θεωρώ ότι εδώ υπάρχουν περιθώρια συνέργειας. Με το Brexit αυτό που θα συμβεί. Ίσως ε, θα έχουμε κάποια παρά, παρόμοια συμφωνία αν έχουμε λοιπόν ευθυγράμμιση Ηνωμένου Βασιλείου από Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό μπλοκ που μπορεί να πιέσει άλλε χώρε. Η Κομισιόν πώ τα βλέπει, Έχει κάποια σχέδια να πιέσει αντίστοιχα κάποιου άλλου εταίρου. Φαντάζεστε ότι καταλαβαίνω, καταλαβαίνετε ε, ότι εννοώ, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι εννοώ, είπα Κίνα και άλλου. Ναι, όμω ο Γενικό Κανονισμό έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την Ιαπωνία, μεν αυτό, ναι, είναι κάπως διαφορετικό, καταλαβαίνω θέλετε να πείτε. Η Άννα. Ε, ε, Βλέπω να υπάρχει στρατηγικό ενδιαφέρον στην αυθυγράμμιση κανόνων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας και να συμμετάσχει και η Ιαπωνία στην προστασία των δεδομένων με την εξέλιξη τεχνολογικών μέσων, την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να έχουμε υπόψη τι αντίκτυπος θα υπάρχει και σε σχέση με το GDPR. Και όταν πήγα στην Ιαπωνία, ασχολήθηκα με τις μεγάλες εταιρείες και τις εξελίξεις τους ε, στο τομέα αυτό. Γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες του GDPR και φροντίζουν να τις εφαρμόζουν. Όμως, το βασικό ερώτημα το είπατε και εσείς πρόεδρε και η Μπυρκίτ. Το θέμα είναι να μην εφαρμοστούν οι κανόνες ε, από την Ιαπωνία προς τους Ευρωπαίου πολίτες, ε, να εφαρμοστούν ε, και στους Ιάπωνες σε ένα βαθμό. Δηλαδή ξέρουμε ότι η αρμόδια αρχή στην Ιαπωνία έχει μια πράξη ανάλογη της του GDPR, αλλά είναι σημαντικό και τα δεδομένα των πολιτών μας στην Ιαπωνία να χρήζουν παρόμοιες μεταχείρισεις. Και κάτι ακόμα. Κάτι που με ενόχλησε και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η, η Ιαπωνία επιτρέπει τα κρυπτονομίσματα και την όλη τεχνολογία που επιτρέπει την άνθηση των κρυπτονομισμάτων να την καλλιεργεί. Τα κρυπτονομίσματα αυτά λοιπόν, ε, μερικά από τα οποία έχουν επενοηθεί από κάποιους που διεκδικούν και την Ιαπωνική ηθαγένεια, ε, κυκλοφορούν χωρίς έλεγχο. Έχω ζήσει στην Ιαπωνία και γνωρίζω πόσο έλεγχο περνάει ε, η κοινωνία της ε, Ιαπωνίας. Ξέρω ότι οι κανόνες εκεί είναι σκληροί. Και καταλαβαίνουμε πώς θα γίνουν σκληρότεροι με την υιοθέτηση της ε, ειδική αυτής πιστοτικής που περιέχει όλα τα στοιχεία των πολιτών. Πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε συμβατοί εάν επιτρέπονται τα κρυπτονομίσματα ε, στην επωνία όπως γίνεται τώρα. Δεν φαντάζομαι τα κρυπτονομίσματα να υπάρχουν χωρί κάποιο είδου παρασκηνιακό τουλάχιστον ή υπόγειο έλεγχο. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Άλλο κανεί. Κύριε Κορέλη. Τζενκαρέλη. Ε, ευχαριστώ. Σε μερικές ερωτήσεις πρέπει να απαντήσω κι εγώ. Αυτή η συζήτηση, αυτός ο διάλογος διαφέρει καθόλου από συζητήσεις και επικοινωνία που έχουμε με άλλες εθνικές αρχές. Η, η μετάφραση των κανόνων που μας δόθηκε από τις Ιαπωνικές αρχές παρόλο που η μόνη επίσημη εκδοχή είναι η Ιαπωνική στο πρωτότυπο, είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας για να μπορέσει κανείς να ξεκινήσει τις συζητήσεις. Η Ιαπωνική αρχή κοιτάζει να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την προστασία που παρέχει. Και βεβαίως, όταν διαπραγματευτήκαμε με τους Ιάπωνες, γιατί οι διαπραγματεύσεις έγιναν ε, στα αγγλικά και μετά μεταφράστηκαν στα ιαπωνικά, μετά κοιτάζαμε να χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουμε, τι εσωτερικέ ε, ειδικέ γνώσει. Έχουμε βεβαίω ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Με υψηλό επίπεδο ε, εμπειρογνωμοσύνη από του ειδικού μα. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε και για το νόημα του κειμένου. Ε, ζητήσαμε βέβαια διευκρινήσεις ε, τα είδαν όλοι οι γλωσσικοί μας ειδικοί, αλλά και ανεξάρτητοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί. Κοιτάξαμε δηλαδή να βελτιώσουμε την κατανόησή μας του Ιαπωνέζικου συστήματος και να μην ε, επαφιόμαστε μόνο σε μία πηγή. Αυτό μας έδωσε την ε, διαβεβαίωση ότι η δουλειά μας στα έγγραφα, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα του επιχάρτου νόμου, είναι το θέμα και της καλής κατανόησης του πώς λειτουργεί το Ιαπωνέζικο σύστημα. Ως προς τα υπόλοιπα ερωτήματα για τους επιπλέον κανόνες. Είναι υποχρεωτικοί και ε, εφαρμόζονται γιατί έχουν βάση στην Ιαπωνική νομοθεσία. Το άρθρο 6 της βασικής πράξης για την ιδιωτικότητα ε, εκχωρεί στην αρχή προστασίας ε, των δεδομένων της Ιαπωνίας επιπλέον δυνατότητες προστασίας, ακόμη και το να χειρίζεται τις διεθνείς ζωέ δεδομένων. Υπάρχει λοιπόν μια κατεξουσιοδότηση, αν θέλετε, πράξη, εφαρμοστική πράξη που επιτρέπει να λάβουν δράση. Οι κανόνες αυτοί είναι και υποχρεωτικοί και ε, άμεσα επιβαλλόμενοι. Χρειάστηκε βέβαια να διευκρινίσουμε κάποιες έννοιες όπως τα ευαίσθητα δεδομένα. Εκεί υπήρξαν κάποιες διορθώσεις όταν μιλούσαμε για μεταφορές δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Προεδρείο, ο Φορέας τη κυβέρνηση, όπου συμμετέχει και ο Υπουργό δηλαδή, για την προστασία των δεδομένων, εκεί εκχωρήθηκαν επιπλέον αρμοδιότητε στην αρχή υποστασία των δεδομένων για να επιβληθούν αυτοί οι πρόσθετοι κανόνε. Η αντιπροσωπεία μα εξήγησε ότι οι κανόνε αυτοί είναι και αυτοί ε, αυστηροί και επιβαλλόμενοι. Οι κανόνε που έχουμε λοιπόν εδώ ταιριάζουν πλήρω στο νομικό πλαίσιο τη Ιαπωνία. Μετά μου θέσατε μια ερώτηση που το βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί οι κανόνες αυτοί, μερικοί από αυτούς, ισχύουν μόνον για τα δεδομένα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επιλογή της Ιαπωνικής Αρχής. Εμείς ως προς το τεστ συμμόρφωσης με τον GDPR, συμβατότητα δηλαδή, μπορούσαμε να ασχοληθούμε μόνο με τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών, των, ε, αυτό που προέρχονται από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι αυτό που ε, οφείλουμε απλώς να κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε, είναι και αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την Ιαπωνική κυβέρνηση, το Ιαπωνικό Κοινοβούλιο. Αυτό που απαιτούν τα ΣΡΕΜΣ και η, το GDPR είναι να υπάρχει αντιστοιχεία. Έτσι κρίνεται η συμβατότητα και να μεταφέρονται μόνο δεδομένα που μπορούν να μεταφερθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό διασφαλίζουν οι επιπλέον κανόνες. Τώρα το εάν λόγω πρακτικών αναγκών οι Ιαπωνικέ εταιρείε θέλουν να εφαρμόσουν δύο διαφορετικά σύνολα ενότητε προστασία των δεδομένων ή επιλέγουν το επίπεδο προστασία συνολικά για όλου, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό το αποφασίζει η Ιαπωνική κοινωνία και οι Ιαπωνικοί θεσμοί. Αυτό που προέχει είναι ότι τα δεδομένα που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε ανάλογο επίπεδο ελέγχου προστασίας δηλαδή. Ως προς τα πρόστιμα. Αυτά τα ποσά προβλέπει από την κοινομοθεσία, αλλά μην ξεχνάμε ότι αφορούν κάθε παραβίαση ξεχωριστά. Είναι αναπαραβίαση. Εάν υπάρξει αδίκημα παραβίαση, θέμα πρόσβαση στα δεδομένα, ε, παράτυπη παράνομη κατοχή δεδομένων που αφορά μεγάλα σύνολα δεδομένων, ιδίω στην ψηφιακή οικονομία, τα ποσά αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν αναλόγως με τον αριθμό των υποθέσεων που συμπεριλαμβάνουν. Και αυτά μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά ποσά. Να τονίσω εδώ ότι πρόκειται για σύστημα διαφορετικό Μιλάμε για ένα ε, δίπεδο, ένα σύστημα με δύο επίπεδα. Κάποια δεδομένα εφόσον είναι παράτημα ή παράνομα και διαγράφονται. Αλλά εάν κάποιο δεν συμμορφώνεται συστηματικά, μπορεί να το επιβληθούν και ποινικές, να ασκηθούν εναντίον του ποινικέ διώξει. Είναι άλλη μορφή κύρωση αυτή τιμωρία από ό,τι προβλέπετε. Συνολικά πάντως, Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πραγματικές κυρώσεις. Και αν δείτε και το τι λέει το Σώμα των Ευρωπαίων Ελεγκτών, δεν πάμε να κοιτάξουμε αν υπάρχει σε μία προσημείο και κεραία προς κεραία ε, αντιστοιχεία στα συστήματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πραγματικές κυρώσεις. Και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να ε, ε, ε, ασκούνται τα ένδικα μέσα και να βεβαιωθούμε ότι το Ιαπωνικό σύστημα λειτουργεί όπως θέλουμε. Και πραγματικά είναι αποτελεσματικό και έχει αποτρεπτικές ποινές. Συμφωνώ απολύτως, η απόφαση αυτή έχει αντίκτυπο πέραν των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι μέρος του ΩΣΑ, του G7, του G20. Έχουμε παρόμοιες ιδεολογικές προσεγγίσεις και για την προστασία των δεδομένων. Η απόφαση λοιπόν αυτή έχει γνωστοποιηθεί στον υπόλοιπο κόσμο. Εάν συγκλίνουμε και στην προστασία των δεδομένων, υπάρχουν άμεσα ωφέλη και για του πολίτε και για τι εταιρείε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντικότατη διάσταση τη όλη υπόθεση. Και για να συνοψίσω για την τελευταία ερώτηση. Είναι επίση πολύ σημαντική απόφαση, μάλλον διάσταση αυτή τη σχέση προστασία δεδομένων Ευρωπαϊκή Ένωση-Ιαπωνία η άλλη σημαντική λοιπόν διάσταση είναι ότι υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ της ιαπωνικής αρχής προστασίας δεδομένων και των δικών μας αρχών προστασίας δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί και μια απόφαση για να υπάρξουν και κοινοί κανόνες ως προς την ερμηνεία και τις νέες εξελίξεις όπως ας πούμε την ε, περίπτωση του blockchain και αυτών των ε, κρυπτονομισμάτων. Και μόλις ληφθεί η απόφαση περί συμβατότητας θα πρέπει να δούμε και τις δικές μας αρχές προστασίας δεδομένων, όχι μόνο ανά επιμέρους υπόθεση, αλλά και το πώς στηρούνται οι κανόνες. Έτσι θα έχουμε περισσότερη νομική προστασία και βεβαιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι απήντησα σε όλα. Όχι, ήσασταν διεξοδικότατος, τι να πω τώρα. Ε, ναι, αλλά δεν αναφέρατε το τελευταίο. Όχι, όχι, δεν με πειράζει. Ε, το χρονοδιάγραμμα, βεβαίω, όλοι έχουμε πρόγραμμα, ακόμη και αυτή η συνεδρίαση που βρισκόμαστε τώρα. Όντω, δύο πράγματα. Ε, υπάρχουν ε, δύο παράλληλες διαδικασίες, αν θέλετε. Οι Ιαπωνικές αρχές πρέπει να ακολουθήσουν τη δική τους διαδικασία για την ε, απόφαση συμβατότητας και αυτό μας έχουν εγγυηθεί ότι θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Και εμείς έχουμε περίπου το ίδιο χρονικό περιθώριο. Βεβαίω θα βιαστούμε αν μπορούμε λίγο, αλλά όχι πολύ γιατί πρέπει να περιμένουμε και την γνωμοδότηση του EDPP. Αλλά όπως είπαν ο πρόεδρος Γιούνκερ και ο πρωθυπουργό Άμπε, στοχεύουμε η απόφαση συμβατότητας να έχει εγκριθεί ως το τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι περίπου χρονικός ορίζοντας, αναλόγως με τα επιμέρους βήματα που θα πρέπει να γίνουν. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τζενκαρέλη και όσοι δεν για όσους δεν πήγαν στην αντιπροσωπεία ή δεν παρακολουθούν το θέμα, όλα αυτά μπορεί να φαίνονται περίεργα και δύσκολα, αλλά είναι βεβαίω πολύ συναρπαστικά και σημαντικά και για την εμπορική συμφωνία και δείχνει ακριβώς πόσο σημαντική είναι η Επιτροπή μας ε, για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Έχουμε δύο λεπτάκια θα περάσουμε σε λίγο στις ψηφοφορίες.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 Λοιπόν, συνάδελφοι, γνωρίζω ότι είστε πολύ άσχολοι την Πέμπτη, να πάρετε και τις πτήσεις και τα λοιπά. Βλέπω ότι έχουμε την ε, απαραίτητη παρτία. Okay, colleagues, let's begin. Um, so the first uh, order of business within the voting. Λοιπόν, το πρώτο θέμα της ψηφοφορίας είναι εκλογή τρίτου αντιπροέδρου για να αντικαταστήσουμε τον Γιάννη Φίλιπ Άρντρεχτ σύμφωνα με το άρθρο 204 του κανονισμού. Λοιπόν, παρακαλώ να έχετε τις κάρτες σας ε, ψηφοφορίας έτοιμες, αλλιώς αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος θα εκλεγεί διαβοής. Σύμφωνα με το άρθρο 200, ανακοινώνω ότι θα έχουμε επίσης τον κύριο Φερχόιν, τον κύριο Κιουτσούκ από την Άλντε και, την κυρία Μύρ του ΙΕΝΕΦ. E Αυτή, είναι τα αναπληρωματικά μέλη. Επίση, οι πολιτικέ ομάδε πρέπει να ενημερώσουν τον Πρόεδρο για αλλαγέ σε αυτόν τον κατάλογο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Για την απαρτία έχουμε περισσότερους από 15 βουλευτές, οπότε έχουμε απαρτία. Ωραία. Λοιπόν, υποψηφιότητες. Παρακαλώ να υποβληθούν υποψηφιότητες για την θέση του τρίτου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Μπορεί να οριστεί υποψηφίος είτε από πολιτική ομάδα είτε από τουλάχιστον 5% των μελών της Επιτροπής, το οποίο σημαίνει τρεις βουλευτές. Μην το κάνετε αυτό σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ αυτό το, τον θόρυβο. Ε, συγγνώμη πρέπει να είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής ε, ο ή υποψήφιος ε, και να έχει υποβάλει δήλωση οικονομικών σφαιρόντων. Πολύ σημαντικό αυτό. Να ε, ρωτήσω λοιπόν ποιοι είναι οι υποψήφοι. Ποιον θέλετε να προτείνετε κυρία Βαλέρο. Την συνάδελφό μου, την κυρία Σαρτζεντίνη. Κυρία Σαρτζεντίνη, λοιπόν, υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Οπότε, να ρωτήσω την κυρία Σατζεντίνη αν συμφωνεί με την υποψηφιότητα αυτή. Θα ήταν τιμή μου, κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ, Τζούντιθ, ε, και τιμή μας η υποψηφιότητά σου. Λοιπόν, τα έγγραφα είναι εντάξει, τα έχει ελέγξει η γραμματεία και πρέπει να τα πω όλα αυτά, έτσι αλλιώς δεν θα είναι σωστή εκλογή. Λοιπόν, όλοι οι υποψήφοι πληρούν τους απαραίτητους όρους, την δήλωση οικονομικών συμφερόντων ε, και είστε τακτικό μέλος της Επιτροπής. Οπότε προχωράμε, επειδή υπάρχει μία υποψήφια μόνο, σε εκλογή διαβοής. Με την άδειά σας, αγαπητοί συνάδελφοι, και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορούμε να περάσουμε στην εκλογή της κυρίας ε, Σαρτζεντίνη ως ε, τρίτης αντιπροέδρου. Διαβοής. Ευχαριστώ. in the future can at least... Και στο μέλλον μπορεί κάποιος άλλος αντιπρόεδρος να βρίσκεται στο Προεδρείο. Δεν ξέρω τι σας έχω κάνει δηλαδή. Δεν δε να κάθεστε δίπλα μου. Δεν είμαι τόσο κακός. Ναι, κυρία Γκάλ, ε, και εσείς ε, ε, ποτέ δεν έρχεστε να καθίσετε εδώ δίπλα μου. Ίσως η κυρία Σαρτζεντίνη να αλλάξει τη συνήθεια. Λοιπόν, επίση λέει στις σημειώσει εδώ πρέπει να πω εκλέγεται η υποψήφια και παρακαλείται να λάβει την θέση της στο Προεδρείο. Να, μα το ήξερα, ορίστε, επιτέλους. Επιτέλους. Πρώτη και τελευταία φορά φαντάζομαι, γιατί κανένας δεν θέλει να έρθει να κάθεται εδώ πάνω αλλά πάντα υπάρχει λοιπόν η θέση σας εδώ όλων των αντιπρόεδρων εάν θέλετε λοιπόν περνάμε στις ψηφοφορίες ναι ναι ε, λίμπε είναι τρέχουμε περνάμε σε επόμενες ψηφοφορίες Has she got the right nameplate? Can you give her a nameplate? Yeah, die heb ik meegenomen. Ja, ja, ja, ja. Okay. Okay, thank you. Congratulations, Judith. Okay, now let's proceed to... Συγχαρητήρια και περνάμε στις ψηφοφορίες. Σημείο 7, 8, 9, 10 και 11 όλες οι συμφωνίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορες χώρες για την απαλλαγή βίζας για σύντομη διαμονή. Ξεκινάμε με την πρώτη. Ο κύριος Εμιλιάν Πάβελ είναι ο εισηγητής για όλες. Ε, θέλει τον λόγο? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τις εκθέσεις αυτές. Ξεκινάμε με την πρώτη. Ε, νέες τροπολογίες αφορά τις ε, νήσες, της νήσους Μπαρμπέιντος. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Ε, what is closed and, the, and that is carried. Δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα τον Μαυρίκιο. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή και αυτή. Σεν Κίτς εν Νέβης. Πέρας. And that is carried. Ε, δεκτή. δεκτή. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή και αυτή. Σε ηχέλες. Και πέρας. Δεκτή. Και τέλος η Συνομοσπονδία των Μπαχαμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και γίνεται δεκτή και συγχαρητήρια στον κύριο Πάβελ και τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Um, και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 13 τη Μαρισιάς διάταξη. Είναι εδώ η συγκεκριμένη κυρία Βίκστρομ. Όποιος δεν θέλει να παραστεί, παρακαλώ να αποχωρήσει ησύχως. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 13, κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Θα ακούσουμε παρουσίαση από την Σεσίλια Βίξτρομ που έχει ετοιμάσει το σχέδιο έκθεσης. Παρακαλώ. Είπαμε λοιπόν κοινωτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και την προστασία. Πολλές επιπτώσεις. Θα τα πει και η κυρία Βίξτον, φαντάζομαι. Έχουμε και κάποιου σκιώδε εδώ. Η Σεσίλη όμω πρώτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που για αλλαγή ανέλαβα κάτι τεχνικό, όχι πολιτικό ή συναισθηματικά φορτισμένο άρα πολύ λιγότερο δραματικό και αμφιλεγόμενο από ε, φακέλους από τον οποίο εργάζομαι συνήθως. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα σημαντικό θέμα. Ποια είναι, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε στο βαθμό του δυνατό θα πρέπει να βασίζονται στην έρευνα, στα ε, στοιχεία. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε καλές πληροφορίες, αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε και τις ορθές πολιτικές αποφάσεις. ένα τομέα όπως αυτό της μετανάστευση ιδίω, που υπάρχουν πολλές πολιτικές διαφωνίες. Πολύ σημαντικότερο σε αυτό το τομέα, λοιπόν, ίσως από άλλους τομείς το θέμα αυτό. Στην έκθεσή μου προσπάθησα να προτείνω νέα θέματα, νέες αποδομαδοποιήσεις στοιχεία που θα πρέπει να παρέχουν τα κράτη-μέλη στη Eurostat. Στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε είτε για στατιστικές που έχουν ήδη ε, εθελοντικά συλλέγουν τα κράτη-μέλη και πρέπει να τις δίνουν στον νέο ζωή κατόπιν τίματο ε, σε φορείς κοινωνίας των πολιτών. Αυτό συμβαίνει ήδη. Αυτό που ζητούμε ίσως ε, αυξήσει τη δουλειά των στατιστικολόγων στα κράτη-μέλη, αλλά είναι σημαντικό νομίζω να μην περιοριστεί η πρόσβαση στις ποιοτικέ στατιστικές λόγω επιχειρημάτων έλλειψης πόρων για τις στατιστικές υπηρεσίες. Αντίθετα πρέπει να έχουν μέσα και κονδύλια οι στατιστικές υπηρεσίες για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους δεδομένου το που δαπανώνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Το πρόσθετο κόστος ε, θα είναι πραγματικά ε, περιθωριακό στο θέμα των στατιστικών. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα. Και ακριβώς η μεγαλύτερη ποιότητα αντισταθμίζει το πρόσθετο κόστος και είπα και ότι θα είναι και ελάχιστο αυτό το κόστος γιατί τα κράτη-μέλη σε πολύ μεγάλο βαθμό με τους πόρους και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους ήδη παρέχουν τα περισσότερα από αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Βεβαίως θα περιμένω να ακούσω τους συναδέλφους και αργότερα να λάβω τροπολογίες. με κατάσταση τροπολογιών είναι η 4η Οκτωβρίου. 5 το απόγευμα. Θέλω να εργαστώ με γρήγορου ρυθμού μαζί με του σκιώδε όταν θα λάβουμε τι ε, τροπολογίε, θα συζητήσουμε μεταξύ μα και ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει πριν το τέλος της θητείας. Και σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο προχωράει γρήγορα και καλά και από ό,τι φαίνεται ούτε και εκεί υπάρχει δυσκολία. Έχουν αντιληφθεί ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων ότι η σημασία των στατιστικών είναι μεγάλη αν θέλει κανείς να πάρει σωστές αποφάσεις έρευνα επιστημονική και αποφάσεις βάσει των αποδείξεων. Σημείωσα την ανακούφισή σου, ε, Σεσίλια, ε, που εργάζεσαι για ένα θέμα που φαίνεται να σημειώνει πρόοδο στον τομέα τη μετανάστευση και ασύλου. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι κανένα θέμα, όσο και αν το λες τεχνικό, οι στατιστικέ δεν στερείται δράματος. Σκιώδης. Η Μαρή Κριστίν, ξέρω, ήθελα να πάρει το λόγο. Εκ μέρους της Γκουε. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν είναι αμυγό τεχνική η έκθεση, αλλά έτσι την παρουσιάστηκε. Το θέμα των στατιστικών είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να εργαστούμε πάνω σε ρεαλιστικά στοιχεία για τις μεταναστευτικές πολιτικές. Και δυστυχώς πρέπει να προοδεύσουμε στη στατιστική για να μην κυνηγάμε φαντάσματα και να είμαστε βασισμένοι σε πραγματικά στοιχεία όσον αφορά τη μετανάστευση. Η Κομισιόν ε, για την ε, παρουσίαση της τροποποίησης κανονισμού λέει ότι αυτό γίνεται για να υπάρξει πασαρμογή στις βαθιές αλλαγές ε, στη μετανάστευση. Εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι ε, να γίνει αυτό ώστε να μπορούν οι πολιτικοί να στηρίζονται σε ρεαλιστικά στοιχεία για να λαμβάνουν σωστέ αποφάσει. Το φάκελο αυτό είναι τεχνικό στη φύση του. Το Συμβούλιο πολύ γρήγορα συμφώνησε. Ελπίζουμε λοιπόν να συμβεί το ίδιο και σε άλλα θέματα. Σε σύλλη αγαπητή, ελπίζω και στο δικό σου θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά όμως γιατί δεν προχωράει τόσο γρήγορα το Συμβούλιο γενικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχει ήδη κάνει, θέλω να σε ευχαριστήσω για την έκθεσή σου, συμφωνώ σχεδόν με όλα ε, όσα προτείνει ε, και με τις προτάσει σου λέω συγκεκριμένα, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη η Eurostat να έχει τα κατάλληλα μέσα. Αφού πρέπει να κάνει πιο πολλή δουλειά, πρέπει να έχει πιο πολλά μέσα στη διάθεσή τη. Η εναρμόνιση δεδομένων είναι μια από τι αρχέ. Υπάρχουν υπάρχει αμφισβήτηση των στοιχείων της Eurostat σε κάθε ε, κράτος. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν μου επιτρέπεις θα πρόσθετα κάποιες προτάσεις και εγώ, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ανήλικους. Πρέπει να είμαστε αρκετά συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά τους ανήλικους ποιες είναι οι πολιτικές επιστροφής, ιδίως εθελούσιας επιστροφής ή μη. Θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις από αυτού. Επίσης, για τον προσδιορισμό της ηλικίας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το διατυπώναμε, αλλά σε πολλές χώρες υπάρχουν προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους που ε, τους ενηλικιώνουν, αν μπορώ να το πω έτσι, τους ε, δηλώνουν ως ενήλικους ή δηλώνονται μόνοι τους ως ενήλικοι. Και επίσης το θέμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Να είχαμε κάποια στοιχεία ε, στο και λίγα για αυτό το θέμα θα ήταν καλό και τα δικαιώματα δηλαδή. Δεν θέλω να παρατείνουμε τη συζήτηση αφού δεν υπάρχει διαφωνία. Έχω και μια ερώτηση προς την Κομισιόν όμως που μας ε, διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει τροποποίηση ό,τι έχω την προστασία των δεδομένων. Εγώ θα ήθελα αυτό να είναι σίγουρο. Δεν θα επηρεάσει δηλαδή τα πράγματα. Θέλω να καθυστηχαστώ γι' αυτό. Αν δούμε δε πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός προστασία των δεδομένων από τα κράτη-μέλη ορισμένε φορές, έχω τις αμφιβολίες μου για το πώς θα μεταφορθεί στα κράτη-μέλη οδηγία αυτή. Ευχαριστώ Μαρή Κριστίν. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν ζητώ συγγνώμη με τη λάθος σειρά σας πήρα. Λοιπόν, ξεκινάμε τελικά με τον κύριο Τσάκη από το ΕΛΚ και μετά η κυρία Κέγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Ντεχόφσκι είναι εισηγητής του ΕΛΚ αλλά απουσιάζει οπότε μου ζήτησε να παρουσιάσω την θέση του ΕΛΚ. Η κυρία Βίκστρομ Ε, είπε ότι είναι τεχνικό ζήτημα, δεν είναι πολύ συναισθηματικό. Εγώ θεωρώ πράγματι ότι αυτό είναι θετικό. Γιατί είναι σαφές ότι στην ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης ε, χρειαζόμαστε περισσότερους ειδικούς. Ενώ οι συζητήσεις μέχρι τώρα ήταν τελείως συναισθηματικές ε, και πολιτικές, ενώ είναι ένα θέμα τεχνικό, πολιτικό και ε, απαιτείται επαγγελματισμός. Οπότε θεωρούμε ότι πράγματι το ΕΛΚ μπορεί να στηρίξει αυτό το ζήτημα. Από την άλλη, το γεγονός ότι για ένα τέτοιο θέμα μπορούμε να συμφωνήσουμε τόσο γρήγορα σημαίνει ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλα ζητήματα. Οπότε είναι πολύ θετικός ο επαγγελματισμός σας. Υπάρχει πίεση στην ευρωπαϊκή πολιτική. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, επαγγελματικές λύσεις. Ε, ο συναλφος Ντεχόσκι έχει γράψει ακριβώς ε, τα σημεία αυτά τα οποία καλώς ορίζουμε. Ε, βεβαίως έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά το σημαντικό είναι να πούμε ότι ο φέκλος αυτός είναι πολύ θετικός, θα τον στηρίξουμε και οπωσδήποτε θα υποβάλουμε και κάποιες τροπολογίες αυτά και συγχαρητήρια στην Σεσίλια. Ευχαριστώ. Η Σεσίλ Κιέγγε είναι ε, από τους Έχετε τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Κλόντ. Ξεκινήσω κι εγώ ευχαριστώντας ε, την εισηγήτρια για το θέμα αυτό το οποίο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της πρότασης της Κομισιόν, δηλαδή να έχουμε καλύτερη ποιότητα εγκαίρως, αλλά βεβαίως να δούμε και την σημασία των στατιστικών. Είναι εξόχως πολιτικό όμως το θέμα πέρα από τεχνικό γιατί ε, πάρα πολλοί ερμηνεύουν την πραγματικότητα με βάση τα όσα θέλουν και φαντάζονται χωρίς να βασίζονται σε δεδομένα και στατιστικά στοιχεία και ανάλογα με το άτομο και την πολιτική τοποθέτηση ε, διαφέρει και η πραγματικότητα. Ε, είναι λοιπόν ε, θέμα εδώ πέρα αντίληψης ε, και γνώσης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τα στατιστικά δεδομένα που είναι στην διάθεση των κρατών μελών που ξαφνικά γίνονται πιο επιφυλακτικά στο να τα μοιραστούν. Λοιπόν, θα πρέπει ακριβώς να ανταποκριθούμε εδώ πέρα στις απαιτήσεις που υπάρχουν και ακριβώς υπήρχαν κάποιες, κάποια κένα στις ε, προτάσεις Κομισιόν θα περιοριστώ στα βασικά. Οι πιο ευπαθείς ε, κατηγορίες, επίσης ε, η διάσταση του φύλου και ειδικά όσον αφορά επίσης οι διαδικασίες αξιολόγησης της ηλικία του αν είναι κάποιος ενήλικος ή όχι, το θέμα της συνοδείας και της ένταξης και της υποδοχής Οπότε θα υποβάλουμε κάποιες ε, τροπολογίες που κινούνται στην ε, γραμμή της συγγήτριας με στόχο να υποβάλουν περισσότερα δεδομένα τα κράτη-μέλη για να έχουμε ένα συνολικότερο πλαίσιο των πολιτικών κράτησης ε, των κρατών μελών, να ζητήσουμε δεδομένα για τη συχνότητα, τη διάρκεια και τον λόγο της κράτησης, αλλά κυρίως δεδομένα για τις εναλλακτικές της κράτησης που πρέπει να μας απασχολήσουν. Επίσης θα ήταν σημαντικό να έχουμε πιο συνολικά δεδομένα όσον αφορά την υποδοχή και την ένταξη και βεβαίως το θέμα είναι η εφαρμογή της ε, υποδοχής αυτής για να μπορέσουμε ακριβώς να δούμε και το τι γίνεται και με τους ε, επαναπατρισμούς και να μπορέσει να έχει τα σωστά στοιχεία η ΕΑΖΟ. Θα συνεργαστούμε λοιπόν στενά με την εισηγήτρια για να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο το οποίο μας χρειάζεται, όπως και τα δεδομένα αυτά, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε και κάποιες αντιλήψεις που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Thank you, Cecil. Um... Ευχαριστώ, Σεσίλ. Αυτά από τους Κιώδης μια στιγμή υπάρχει μια ερώτηση από την Μαρή Κριστίν προς την Κομισιόν. Σας πειράζει να την ακούσουμε. Αν θέλει η Κομισιόν. Ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σας διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν παρκείς εγγυήσεις στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Δίκαιο που προβλέπουν ακριβώς την διασφάλιση ε, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σεσίλια, θα ολοκληρώσετε. Thank you very much and thanks to all colleagues. Well, Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Ε, χαίρομαι που είμαστε όλοι μια ομάδα ενωμένη και βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η Μαρή Κριστίν έθεσε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Ε, θα το δούμε και θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Επίσης ήμουν σε επαφή και με το Συμβούλιο. Σήμερα ή χτες, νομίζω, κατέληξαν σε μια συμφωνία όπως αντιλαμβάνομαι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό γιατί σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι χρειαζόμαστε στοιχεία αξιόπιστα και εναρμονισμένα αυτό είναι και το αντικείμενο της πρότασής μας ε, και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδελφούς και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Προφανώς ε, είναι πολύ σημαντικά τα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για να μιλάμε με στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Βίκστρομ. Ευχαριστώ συνάδελφε που είστε όλοι εδώ. Ξέρω ότι είναι πέμπτη απόγευμα. Οπότε ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο προβλέπεται για τις 11.30 και επειδή δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι για να πάρουν το λόγο, προτείνω να κάνουμε μια διακοπή μέχρι τις 11.30. Αν μπορείτε να το δεχτείτε, συνάδελφοι, να διακόψουμε. Διότι οι ομιλητές μας για το επόμενο σημείο, του Ιουλίσσα, e θέλουμε να φτάσουν. Uh, happens, which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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Υπότιτλοι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

Sorry, colleagues, for the slightly late start. There's a lot of um, issues going on. This always happens on Thursday. Συνεχίζουμε. Ε, τώρα αυτά συμβαίνουν τις πέμπτες. Τι να λέμε. Σας ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, που ήρθατε, κυρία Τζανίτσι, μόνο εσείς. Και το κρατάμε ανοιχτό το μαγαζί. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, συνάδελφοι από την EU Λίζα και ο Κύριο Γκάρκοφ, ο Γενικός Διευθυντής, ε, εκτελεστικός διευθυντής. Καλώς ήρθατε. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης ε, της υπηρεσίας ε, και περιττό είναι να πούμε ότι έχουμε μια στενή σχέση εργασίας με την υπηρεσία σας. Την τελευταία φάση αυτή της συνεργασίας και της λογοδοσίας η υπηρεσία έχει εφαρμόσει πολλά νομοθετήματα τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Λίμπα και είναι άρα ακόμη σημαντικότερο να ακούσουμε την παρουσίασή σας την σημερινή. Σας συγχαίρω και για τα νέα σας γραφεία στην έδρα σας στο Ταλίν που εγκαινιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα μόλις. Πρέπει να έρθουμε να τα δούμε κάποτε. Ελπίζουμε. Και Γνωρίζω ότι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θα πάνε ή έχουν πάει, δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε Γκάρκοφ, αν μπορείτε να μας κάνετε την παρουσίαση. Ελπίζω να έρθει και κανένας βουλευτής κάποτε, αλλά μεταδίδονται και στο διαδίκτυο. Αυτά, οπότε κάποιος θα παρακολουθεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, ξεκινήστε εσείς κύριε Γκάρκοφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Είναι πάντα ευχαρίστησή μας να ερχόμαστε εδώ και να παρουσιάζουμε τα επιτεύγματα της Υγιού ε, Λίζα. Για το 2017 είχαμε ένα χρόνο δύσκολο αλλά ικανοποιητικό. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια διπλή πρόκληση αφενός να διατηρήσουμε τις τρέχουσες επιχειρήσεις, τα υφιστάμενα συστήματα και ταυτόχρονα να συνεχίσει η συνεισφορά της ε, και να αυξηθεί η συνεισφορά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Συνολικά ε, κλείσαμε πέντε έτη το 2017, ε, μια περίοδος δηλαδή που προσφέρεται για μια ανασκόπηση και οφείλω να πω ότι επιτύχαμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την βελτίωση της παροχής ε, ποιοτικών υπηρεσιών, ε, βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων μεγάλης κλίμακας, αποδεικνύοντας έτσι ότι έχουμε έναν επαγγελματικό φορέα, κάτι το οποίο ήταν η σωστή απόφαση, αποδείχτηκαμε ένας αξιόπιστος και ικανός εταίρος ε, των κρατών μελών και βεβαίως καταφέραμε να αναλάβουμε και νέα καθήκοντα για να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια, την διαχείριση των ε, συνόρων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων μας έχουν εμπιστευτεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και το Eurodac και οφείλω να πω ότι δεν είχαμε κρίσιμα συμβάντα που να αποτρέψουν την φυσιολογική μας λειτουργία. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Στο τέλος του 2017 πάνω από 76 εκατομμύρια συναγερμούς ε, ειδοποιήσεις ε, είχαμε εισαγαγή στο σύστημα. Ο αριθμός αιτήσεων βίζας στο σύστημα βίζας ήταν πάνω από 52 εκατομμύρια και η Eurodac αποθηκεύσε πάνω από 5 εκατομμύρια αρχεία ετούντων άσυλο ή παρατύπων μεταναστών, οπότε υπάρχει μια σαφής ε, τάση ευρύτερης χρήσης ε, του συστήματος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Επίσης, οφείλω να πω ότι τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την ομαλή λειτουργία της περιοχής ε, Σέγγεν και για την σωστή χάραξη πολιτικής ε, ασύλου. Οπότε δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα συστήματα που διαχειρίζεται σήμερα η υπηρεσία μας είναι ο θεμελίος λήθος ε, της πολιτικής αυτής και βέβαια συνεισφέρουν στην εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Οπότε στο μέλλον όσο η κατάλληλη ε, όσο υπάρχει η τρομοκρατική απειλή και η μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα και εξαρτάται από την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσω ευέλικτων και διαλειτουργικών συστημάτων πληροφορικής που θα πρέπει να έχουν οι αστυνομικέ αρχές, οι συνοριοφύλακες ε, και οι αρμόδιοι για τη μετανάστευση. Κάποια περισσότερα στοιχεία με το SIS2, την τεχνική ένταξη της ε, Κροατίας ολοκληρώθηκε, οπότε η Κροατία είναι έτοιμη πλέον να ενταχθεί στην ζώνη Σέγγεν. Επίσης το 2017 ολοκληρώσαμε την ανάπτυξη του συστήματος δακτυλοσκόπησης ε, που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο φέτος. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 κρατη που χρησιμοποιούν το σύστημα και άλλα 4 προετοιμάζονται. Τον Μάιο Είχαμε πάνω από 21.000 αναζητήσεις ε, βιομετρικών δεδομένων ε, και τον Ιούνιο 40.000 αναζητήσεις. Είχαμε σοβαρές ε, εξέλιξεις με το σύστημα πληροφοριών Visa, όπου είχαμε μια νέα αναβάθμιση του συστήματος που προβλέπει τις αλλαγές των κώδικα Visa και ακριβώ ήταν κάτι το περίπλοκο και σημαντικό και βεβαίως θα υπήρχε πρόβλημα με την ασφάλεια της περιοχής Σέγγεν εάν ε, δεν λειτουργούσε, οπότε δεν υπήρχε περιθώριο λάθος. Το έργο όμω ολοκληρώθηκε εγκαίρω και εντό ε, του προπολογισμού. Επίση το 2017, μαζί με τα κράτη-μέλη, η υπηρεσία μα ε, προχώρησε σε μια άσκηση συνέχεια λειτουργία και ανάκτηση από καταστροφή για να δούμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποια ε, καταστροφή και τα αποτελέσματα βεβαίως ε, προωθήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορούμε να χειριστούμε 7 εκατομμύρια αρχεία και 1.200 συναλλαγές ανά ώρα και τον Ιούνιο του 2017 η Europol έλαβε πρόσβαση στην ε, βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και άρχισε να τη χρησιμοποιεί, αλλά η δουλειά της υπηρεσίας μας το 2017 δεν περιορίστηκε μόνο στην καθημερινή ε, δουλειά που κάνουμε αλλά το 2017 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην προετοιμασία του συστήματος εισόδου-εξόδου. Έγιναν οι απαραίτητες προσλήψεις, ξεκίνησαν οι αναγκαίες διαδικασίες προκήρυξης και από κοινού με τα κράτη-μέλη προετοιμάσαμε τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος. Τέλος, ε, δώσαμε σημαντική στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία πράξεων κατεξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 36 του σχετικού κανονισμού που ε, ολοκληρώθηκε έγκαιρος. Επίσης ε, φροντίσαμε να δράσουμε προληπτικά έγιναν οι αρχικές εφαρμογές ε, Παρασκευής ε, επισκέψεις στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και στο Λονδίνο και συζητήσαμε τις σχεδικές τους εμπειρίες όσον αφορά την εφαρμογή των ενιαίων συστημάτων για τις χώρες τους επίσης. Συνεχίσαμε την στήριξή μας σε ζητήματα διαλειτουργικότητα. Συγκεκριμένα δώσαμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για το κοινό βιομετρικό σύστημα και έτσι όλα αυτά αποτέρεσαν την αφετηρία για την περαιτέρω δουλειά στις τεχνικές πτυχές για την προετοιμασία της διαλειτουργικότητας στα επόμενα έτη. Η υπηρεσία επίσης ε, προετοίμασε τον ε, συντονισμό του σχεδίου δράσης για την ποιότητα των ε, δεδομένων και ε, εκεί πέρα βεβαίως συναντήθηκαν διάφορα μέρη που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας, όπως προβλέπει το άρθρο 8 του αναθεωρημένου κανονισμού. Το 2017 η υπηρεσία μας επίσης ε, έκανε πάνω από 40 διαφορετικές εκπαιδεύσεις ε, στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, χρήση του συστήματος και αυτό δεν αφορούσε μόνο τους πληροφορικάριους αλλά και λιποπροσωπικό. Και τέλος, το 2017 η υπηρεσία μας αύξησε τη συνεισφορά της στο μηχανισμό κανονισμού Σέγγεν, όπου οι ειδικοί ήταν ε, παρόντες σε 8 αποστολές αξιολόγησης ε, και ακριβώς ε, στηρίξαμε τις πολιτικές βίζας. εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας, διαχειριστήκαμε έναν προϋπολογισμό 153 ε, εκατομμυρίων δεσμεύσεων και 67 εκατομμυρίων πλήρωμων και σας ενημερώνω ότι τα εξαντλήσαμε σχεδόν στο 100%. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να αναφέρω πως ε, η χρονική καθυστέρηση στην έγκριση των νομοθετημάτων δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην εφαρμογή του προϋπολογισμού και απαιτεί περαιτέρω δράσεις, ε, κατά το οποίο ίσως αργότερα σημάνει δυσκολίες ε, στις διαδικασίες ε, προμηθειών ή αδυναμία να εξαντληθούν οι διαθέσιμες πιστώσεις. Όσον αφορά την στελέχωση, το 2017 είχαμε 167 άτομα προσωπικό 121 προσωρινούς ε, και οι υπόλοιποι ήταν μόνιμο προσωπικό και εθνική αποσπασμένοι υπάλληλοι και προβλέφθηκαν άλλες τέσσερις θέσεις ε, για τον κανονισμό εισόδου-εξόδου. Για το επιτελείο μας, ε, η οικοδόμηση ξεκίνησε το 2017, ολοκληρώθηκε τον Μάιο. η διαδικασία εκμίστοσης Δεν έχουμε ακόμα έδρα στο Τάλιν, απλώς στεγαζόμαστε και στο Στρασβούργο. Η οι υπηρεσίε μα πήγαν στο νέο κτίριο, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι οι χώροι που έχουμε θα είναι αρκετοί για τι νέε αρμοδιότητε του οργανισμού. Χρειαζόμαστε και υπαλλήλου και τα απαραίτητα συστήματα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και τη δεύτερη φάση οικοδόμηση τη προέκταση, που θα καλύψει τι ελλείψει που έχουμε εντοπιστεί. Ο οργανισμός έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις. Δεν θα σας τα διαβάσω τώρα όλα, να αναφέρω τα βασικότερα που αντιμετωπίσαμε. Την επάνδρωση της προσλήψης. Το 2017 ο οργανισμός αναγκάστηκε να φέρει εις πέρα στις αρμοδιότητές της και τις υποχρεώσεις τη με μειωμένο προσωπικό, μειώσεις που προβλέφθηκαν από το 2014. Όντως, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση του υπαλληλικού μας προσωπικού, αλλά παρόλο που αυτό το καλώς ορίζουμε, για να μπορούμε να λειτουργούμε εύρυθμα, Έχουμε τόσε οριζόντιε λειτουργίε που χρειαζόμαστε περισσότεροι επάντρε, περισσότερε προσλήψει. Υπάρχει κίνδυνο να μην φτάσουμε στο επίπεδο των ε, απαιτήσεων για τις αρμοδιότητες που μας έχουν ανατεθεί. Υπό αυτήν την έννοια το 2018 και τα επόμενα χρόνια Ο οργανισμό θα πρέπει να ενισχυθεί το δυνατόν περισσότερο βεβαίω με την ε, Συμφωνία των Ευρωπαϊκών Αρχών. Μιλάμε για οριζόντιε λειτουργίε πέρα από την λειτουργία του ίδιου του οργανισμού. Για να ολοκληρώσω, εμεί ο οργανισμός για την λειτουργία των ψηφιακών συστημάτων στον χώρο ελευθερία δικαιοσύνη και δημοκρατία. Είχαμε μέχρι τώρα επιτυχή αποτελέσματα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και τα ερχόμενα χρόνια ώστε να λειτουργεί ε, σωστά ο χώρο Σέγγεν και να ανταποκρινόμαστε εγκαίρω στι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα συστήματα και οι υπηρεσίε μα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία τη Ένωση. Όπω λέω συχνά, σήμερα είναι γοργά μεταβαλλόμενο ο ψηφιακό κόσμο και απαιτείται για τη διαχείριση της μετανάστευσης και όλων των ε, ειδών κυκλοφορίας. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε με τεχνολογικές λύσεις αξιόπιστες να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερη και δυνατότερη. Ευχαριστούμε κύριε Κέρχοπ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κινίτση και την κυρία Σβιεύτσκα. Θέλω να αφήσω και εγώ μια ερώτηση. Πώς θα συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες που ανακύπτουν μέρα τη μέρα με το διευρυμένο πεδίο αρμοδιοτήτων σας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σχολιάσετε. Γιατί γνωρίζετε καλύτερα εσείς τις δυσκολίες εκ των έσω. Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς το καταλαβαίνω εγώ απ' έξω. Μπορείτε να σχολιάσετε τα προβλήματα διαλειτουργικότητας είναι πολιτικά αμφιλεγόμενο αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερη διαλειτουργικότητα. Εσείς μελετήσατε την πρόταση που υποβλήθηκε ε, πρόσφατα. Πόσα διαδομένα θα μπορείτε να καλύπτετε με τη διαλειτουργικότητα, πώς θα το διαχειρίζεται η, η Γιουλίζα και τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στη διάρθρωση των ψηφιακών συστημάτων οι δυσκολίε που θα έχετε να αντιμετωπίσετε δεν είναι κλασικέ κλασικές του Ιουλίζα, θα είναι καινούργιε και θα είναι σημαντικές. Και επειδή δεν καταλαβαίνουμε τις βάσεις δεδομένων τόσο καλά απ' έξω, Πείτε μας εσείς. Η τεχνολογία φέρνει αλλαγές. Πώς θα αντιμετωπίσει η Γιουλής αυτές τις αλλαγές. Έχετε τα απαραίτητα εργαλεία. Κατερίνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το Διευθυντή Ντάρκοφ για την τόσο κατατοπιστική ομιλία του και τις δραστηριότητες της Λίζας. Πρόσφατα μπόρεσα να επισκεφθώ τον οργανισμό σας και εργάστηκα και του κανονισμού για την αναδιάρθρωση του Λίζα και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που σας περιμένουν για να διαχειριστείτε τι βάσει δεδομένων που είναι όλο και περισσότερε και περίπλοκες. Θα καλύπτονται πλέον και τα συστήματα όπως το έκρης, το αίτιας και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την τόσο λεπτομερή παρουσίαση που κάνατε. Και αν μπορείτε να απαντήσετε και σε κάποιες από τις δικές μου τις ερωτήσεις. Γνωρίζοντας ότι ο οργανισμός η Γιουλίζα έχει ήδη πετύχει σοβαρά αποτελέσματα για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη ως προς την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και τη σωστή διαχείριση των συνόρων για να υπάρχει και η δημόσια ασφάλεια. Ήδη το σχολιάσατε και εν μέρει απαντήσατε σε μια από τις ερωτήσεις μου. Το θέμα της βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων. Αυτό νομίζω ότι είναι μια βασική πτυχή. Όπως επίσης απαντήσατε και στο θέμα της ενημέρωσης, διότι η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και εκπαίδευση, κατάρτιση, είναι αλληλένδετα στοιχεία. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν μπορούμε να ξαναπάμε σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη και τη συνεισφορά του οργανισμού σας, για μια ικανοποιητική εκπαίδευση των υπαλλήλων και κατ' επέκταση αυτών που εργάζονται και στα κράτη-μέλη, ώστε και τα ίδια τα κράτη-μέλη μέσα από αυτό το σύστημα να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα από μόνα του. Έχουν υπάρξει δυσκολίε. Αν έχουν μάλιστα υπάρξει και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, τι λύσει βρήκατε για να τι υπερβείτε. Ιδίω σα προ την εκπαίδευση του προσωπικού σα. Ένα άλλο θέμα που θίξατε και είναι σημαντικότατο είναι αυτό των πόρων. Εάν θυμούμε σωστά, Ο αριθμός των υπαλλήλων σας ήταν ένα από τα λίγα επικριτικά σχόλια που έγιναν στη διαδικασία ε, απαλλαγή που ε, περάσατε πέρσι την ετήσια διαδικασία απαλλαγή. Τώρα μας λέτε ότι χρειάζονται περισσότερες προσλήψεις. Σας ρωτώ, είναι απαραίτητη, είναι ε, επαρκής η επάνδρωση του οργανισμού. Διότι αν πρέπει να πάρετε περισσότερους υπαλλήλους θα χρειαστούν και περισσότερα κονδύλια. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ανάλογη αύξηση. Και αυτό θέλω να σχολιάσετε. Και, ένας, και άλλο ένα ερώτημα γενικό που σχετίζεται και με αυτό που είπε και ο πρόεδρος Μωράης. Μιλήσατε για τη διαλειτουργικότητα. Μιλήσατε για τα βιομετρικά δεδομένα. Εδώ επιβάλλεται το να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή προσοχή στην ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Υπάρχουν οργανισμοί που ασχολούνται ακριβώς με αυτό, όπως ο ΦΡΑ, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Χρειάζεται απαραίτητη διάρθρωση αυτών των οργανισμών. Ερωτώ λοιπόν εάν και με ποιου όρου ο οργανισμό σα, η Γιουλίζα, συνεργάστηκε με αυτού τους οργανισμού ακριβώ για να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη η απέτηση να υπάρχει ο μέγιστος δυνατός ε, βαθμός προστασίας των δεδομένων. Και ολοκληρώνοντας, να ρωτήσω και πώς ο οργανισμός σας συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα. Ώστε τα πρότυπα, τα αυστηρός τεχνικά και τις ασφάλειες να είναι στο δυνατόν υψηλότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να σας ε, συγχαρώ για την πολύ καλή σας δουλειά, κύριε Γκάρκοφ, για το 2017 και κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την ένταξη της Κροατίας ε, στο SES, e την αναθεώρηση και αναβάθμιση στόματος βίζα και το σε το σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Έχω ένα ερώτημα για διαλειτουργικότητα. Γνωρίζω ότι ο οργανισμός στηρίζει τη μελέτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα μέσα διαλειτουργικότητα. Όχι μόνο αυτά τα οποία συζητήσαμε στο πλαίσιο των τριμερών ε, διάλογων για την πρόταση ενίσχυση ε, τη εντολή σα, του οργανισμού σα εννοώ. Τι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Πύλη και στο κοινό αποθετήριο για να αξιοποιούμε το χρόνο μας και την ασφάλεια του συστήματος. Σας ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Κύριε Γκάρκοφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κινίτση και την κυρία Κουρτσκά που έδειξαν ότι εκτιμούν το έργο του οργανισμού μας και θα προσπαθήσω να απαντήσω στο κοινό σας ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα φυσικά και είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Όμως έχει πλέον ε, μπει στο προσκήνιο σε πολύ επικυριχρονική στιγμή όταν πλέον έχουμε επιτύχει μια κρίσιμη μάζα πληροφορικών συστημάτων σε επίπεδο ένωσης και κρατών μελών. Υπάρχει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τον ιστορική ασφάλεια, τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων. Θα πρέπει λοιπόν η τεχνολογία που στόχο έχει εν γέννη την υποστήριξη και τη διευκόλυνση το έργου των συνοριοφυλάκων, τελωνιακών και λοιπόν να είναι κατάλληλη. Και η διελτουργικότητα βοηθάει. Από μόνη της βέβαια η διαλειτουργικότητα δεν δημιουργεί νέες βάσεις δεδομένων, οι ομαδοποιήσεις ή ε, συγχωνεύσεις δεδομένων, όχι. Απλά επιτρέπει τη πιο αποτελεσματική χρήση αυτού που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας σήμερα. Χρειάζεται και διαχείριση πιο αποτελεσματική για τον καθορισμό της ταυτότητας. Και αυτό θα βοηθήσει την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων μαζί με αυτή την προσέγγιση σταγανοποίησης, ε, σιλό. Εμείς συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως όπως μας έχει ζητηθεί στηρίζουμε και τις διαπραγματεύσεις για την πρόταση, παρέχουμε εμπειρογνωμοσύνη και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια επιτυχή συμφωνία σε ό,τι αφορά την πρόταση διελειτουργικότητας τόσο των προσεχών μηνών. Έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να προγραμματίσουμε την πρακτική εφαρμογή των συνιστοσών της διαλειτουργικότητα. Και θα εντάξουμε στην αρχιτεκτονική της δελτουργικότητας στα νέα συστήματα. Αυτό είναι πρόκληση. Όχι μόνο τεχνική για τη διαλειτουργικότητα Είναι τεχνική πρόκληση. Η βασική πρόκληση του οργανισμού μας στον τομέα αυτό είναι οι άλλες πρωτοβουλίες πλην της δελτουργικότητας που θα πρέπει να αναλυφθούν ταυτόχρονα. ταυτόχρονα. εξοδος το προφανές αίτια Θα τεθεί σε ισχύ σύντομα ο κανονισμό αυτός, το είπε και ο πρόεδρο. Έχουμε και αναδιατύπωση νομοθετικών μέσων που διέπουν αυτά τα συστήματα. Είναι σε διαπραγμάτευση ορισμένε αυτές ε, οι ε, τίθενται σε ισχύ. Άρα ε, τρία με πέντε χρόνια ορίζοντα. Καλύπτουμε και αυτές είναι βασικέ μα μας προκλήσεις. Ταυτόχρονα, Όπω κάναμε μέχρι τώρα, έτσι και στο μέλλον θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Με την προπόθεση να έχει οικονομικούς πόρους επαρκής, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό επαρκές η υπηρεσία μας. Ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια των δεδομένων, ήδη σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα συστήματα που διαχειριζόμαστε διακρίνονται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας ε, πρόσβαση, φυσική ασφάλεια δηλαδή, οργανωτικά μέτρα. Άρα, περιορισμένα τα άτομα που έχουν πρόσβαση και μέτρα ασφάλειας κυβερνοχώρου για την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων. Τα ίδια μέτρα, βέβαια, θα εφαρμοστούν και στα νέα συστήματα και στην αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας που θα αναπτυχθεί. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των δεδομένων. Ήδη έχει κάνει πολλά για την ποιότητα των δεδομένων στα συστήματα ο οργανισμός μας. Σας είπα ότι ξεκινήσαμε ήδη από το 2016, συνεχίσαμε το έργο το 2017, κάναμε τακτικές εκθέσεις στα κράτη-μέλη για παρεκκλήσεις από τα τρέχοντα ποιοτικά πρότυπα Βλέπουμε όλο και περισσότερες δράσεις από τα κράτη-μέλη για την διόρθωση των προβλημάτων. Το 2017 ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση σε, τα σε σχέση με τα προηγούμενα έτοιμα και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Περιμένουμε να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμό κανονισμός για να μπορέσουμε να προβούμε στα επόμενα βήματα και αποκοινούμε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσουμε κοινού ποιοτικού δείκτε και πρότυπα που θα εφαρμόσουμε εν συνεχεία στα συστήματα της Ένωσης, αλλά και στα σχετικά εθνικά. Αυτό θα οδηγήσει σε μια σημαντική θετική αλλαγή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων σε σύγκριση με το παρόν. Εκπαίδευση, δημιουργία αποδομών και δυνατοτήτων. Σίγουρα είναι ένα θέμα που πολλές φορές το λησμονούμε, αλλά είναι και πολύ σημαντικό αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα που έχουμε αναπτύξει και όπως είπα το 2017 ο οργανισμός μας ε, έκανε 42 ε, μαθήματα και το χαρτοφυλάκιο θα το επεκτείνουμε και στα επόμενα χρόνια. Έχουμε προκλήσεις γιατί έχουμε ζήτηση όλο και μεγαλύτερα από τα κράτη-μέλη Δηλαδή καταλαβαίνουν όλο και περισσότερο ότι πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη υποδομών και δυνατοτήτων, αλλά δεν έχουμε πόρους να αφιερώσουμε στις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες. Και από πλευρά ανθρώπινων δυναμικών έχουμε μόνο έναν υπεύθυνο εκπαίδευση. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Προσλαμβάνουμε εθνικού εμπειρογνώμονε. Δεν πετυχαίνει πάντα αυτό βέβαια, γιατί δεν θέλουν και τόσο πολλοί εθνικέ διοικήσει να μα στείλουν τους καλύτερους ε, δυνατούς εμπειρογνώμονες, αλλά με την ενίσχυση που προβλέπετε και αυτήν και μια από τις που σας έλεγα πριν, ελπίζουμε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Με τη στήριξη ιδίω της ε, Δημοσιονομικής Αρχής. Εκπαίδευση στα κρατημέλη. παρέχουμε μαθήματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Να δημιουργηθούν εσωτερικές δυνατότητες και υποδομές για να μπορούν οι τελικοί χρήστες να εκπαιδεύονται στις χώρες μέλη. Επίσης, προλαμβάνουμε, προβλέπουμε τις ανάγκες που θα προκύψουν από τα νέα συστήματα αίτιας, σύστημα εισόδου-εξόδου, ΣΕΠΟΛ και Frontex. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις δύο υπηρεσίες. Θα φτιάξουμε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα σπουδών ή εκπαίδευσης και το 2019 θα αναπτύξουμε το πακέτο, το χαρτοφυλάκι όλων αυτών των μαθημάτων που θα αρχίσει να εφαρμόζεται, να παρέχονται δηλαδή αυτά τα μαθήματα από το 2020-2021. Άρα αντιδράμε εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Διαλειτουργικότητα ζέων θέμα στο πλαίσιο της προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή. Απαντώντας σε ένα από τα ερωτήματα του Προέδρου. Η διαλειτουργικότητα δεν θα δημιουργήσει από μόνη νέα συστήματα. Άρα δεν χρειάζεται να προστατευτούν νέα συστήματα ή νέα δεδομένα. Η ίδια προστασία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και με την νέα αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητα. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται. Πρέπει όμω να γίνει διάκριση μεταξύ ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων. Η προστασία δεδομένων σημαίνει πώ προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα και αυτό είναι ευθύνη του οργανισμού. Και βέβαια ο επόπτης δεδομένων μας εποπτεύει. Δεν υπήρξε αυτά τα πέντε χρόνια κάποια κριτική μετά από τις επιθεωρήσεις που έκανε ο Ευρωπαϊκός Επόπτης. Η ιδιωτικότητα αφορά πιο πολύ τον τρόπο χρήση του συστήματο. Άρα ευθύνη εδώ, την ευθύνη την έχουν τα κράτη-μέλη. Ιδίω μιλώ για τα νέα συστήματα. Privacy by design είναι ο κανόνας. Αυτή είναι η αρχή που εφαρμόζουμε. Και βέβαια συνεργαζόμαστε με τον Οργανισμό Θεμελιών Δικαιωμάτων, και λάβαμε υπόψη την πρόσφατη έκθεση τους ε, για την χρήση των, ε, και τη λειτουργία των συστημάτων ε, πληροφορικής μεγάλης κλίμακας. Θα λάβουμε υπόψη τις συστάσεις του. Και για το σχεδισμό του αίτιας. Τέλος, συντονισμός με τον ιδιωτικό τομέα. Από την αρχή που ιδρύθηκε ο οργανισμός, εστιάσαμε σε ανοιχτές εταιρικέ σχέσεις με του διαφορού εταίρου. Είμαστε τεχνολογικό φορέα, αλλά δεν είμαστε αυτοί που καινοτομούμε, ιδιωτικό τομέα καινοτομεί. Και εμεί πρέπει να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νέα χαρακτηριστικά και τι νέε τεχνολογίε υπέρ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Η καλή πρακτική που έχουμε είναι η διοργάνωση αιτήσεων, εκδηλώσεων, διασκέψεων, στρογγυλών τραπεζιών για τη βιομηχανία και εκεί εξετάζουμε διάφορα στήματα. Τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, το θέμα μας θα είναι τεχνολογία και πώς εφαρμόζεται στα εξωτερικά σύνορα, τα χερσαία εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για να διευκολύνει τη χρήση των συστημάτων εισόδου-εξόδου και του αίτιας. Έχουμε οικοδόμηση μια πολύ καλή σχέση αυτή την πεντέτεια με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίω αυτούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, σωματικότερους παίκτε. Ε, και το 2015 είχαμε ενεργήσει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα και είδαμε και τι έχει γίνει μέχρι τώρα την κυρία Διατουρικότητα, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει με το SPN, CR, για τη διατήρηση ασφάλειας. Και τα δύο στοιχεία ισχύουν. Δεν κάτι καινούριο. Και χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόσβαση στα δεδομένα. Να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Οι ίδιοι κανόνες πρόσβασης που τώρα ισχύουν για τα συστήματα Eurodac κτλ. θα χρησιμοποιηθούν για το ESP και Έτσι θα αγγιθούμε την αρχή της, του περιορισμού των, της πρόσβασης. Δεν θα αλλάξει η χρήση των δεδομένων σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Τα μεμονωμένα συστήματα χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα. Απλά θα έχουμε πολύ πιο αποτελεσματική πρόσβαση. Άρα θα έχουμε ωφέλη για τι αρχέ διαχείριση ε, συνόρων επιβολής νομοθεσίας, μετανάστευση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ και ελπίζω ότι κάλυψα όλε τι ερωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και στους δύο συναδέλφους που ήρθαν. Κύριε Γκερκόφ, χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε και θα σας δούμε πάλι σύντομα. Τελειώνουμε με την πρωινή συνεδρίαση. Έχουμε στις 12.30 τους συντονιστές και μετά θα ξαναρχίσουμε στις 3. Η ακρόαση για την οδηγία 13.30. Καλή όρεξη συνάδελφοι. coordinators in this room.